La séance est reprise. Συνεχίζεται η συνεδρίαση. Nous reprenons la séquence des Συνεχίζουμε λοιπόν με ψηφοφορίες και πρέπει να ψηφίσουμε για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, EUOSHA, ε, ε, γνωμοδότηση του κυρίου Γκάιερ. Έχουμε αρκετές τροπολογίες και θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Μοντέλ, τη συνάδελφό μας, η οποία εργάστηκε πολύ εντατικά, που θέλει να μεταφερθεί η υπηρεσία αυτή που βρίσκεται στην Ισπανία και να πάει στην Μπουρκόνη. Δεν ξέρω αν ο Δούκας της Βουργόνης μπορεί να είχε κυριαρχία στην Ισπανία, αλλά δεν ξέρω εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ε, μα μας ε, μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Επομένως, η τροπολογία 243 είναι μη παραδεκτή. Πρώτη τροπολογία, τροπολογία 26 στο άρθρο 1. Έχει ε, λογική η οποία συνάδει με άλλες τροπολογίες και θέλουμε εδώ να ομοδοποιήσουμε unblock τις ε, τροπολογίες διαγραφής για τα διάφορα άρθρα. Η τελική λογική είναι να καταργηθεί ο οργανισμός. Εάν λοιπόν υπάρξει πλειοψηφία υπέρ κατάργησης του οργανισμού θα κερδίσουμε και χρόνο. Προτείνω όμως να ψηφίσουμε unblock όλες τις τροπολογίες οι οποίες επιθυμούν διαγραφή ε, άρθρου γιατί ούτως ή άλλως ο στόχος είναι κοινό και μετά θα δούμε από εκεί και πέρα τις τροπολογίες που αφορούν τις διάφορες παραγράφους και ε, τις διάφορες περιπτώσεις θα τις δούμε ε, αναπερίπτωση αλλά επειδή ε, εδώ είμαστε πάντα προς την ίδια κατεύθυνση και θα δούμε την άποψη της Επιτροπής. Προτείνουμε λοιπόν να ψηφίσουμε μπλοκ για όλες τις τροπολογίες οι οποίες αφορούν ε, άρθρα διαγραφής. Εάν θέλετε λοιπόν να διαγράψετε τα διάφορα άρθρα, σας παρακαλώ σηκώστε το χέρι σας. Αν δεν θέλετε να διαγραφούν τα άρθρα τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Κατά. Αποχές δεν βλέπω κανέναν. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλες οι τροπολογίες οι οποίες ζητούν διαγραφή οποιοδήποτε άρθρου απορρίπτονται. Τροπολογία 29 του κυρίου Νεγκρέσκου αποσύρεται. Τροπολογία 31 της κυρίας Μοντέλ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 32 και πάλι διαγραφής υπέρ, κατά, αποχής, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται.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 55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 αποσύρεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ποιος θέλει το λόγο? Ο κύριος Φερνάντες. Βλέπω ότι ένα συνάδελφο ζητά συνέχεια την ίδια ε, τροπολογία διαγραφή-διαγραφή. Προτείνω οι τροπολογίε της κυρία Μοντέλ που είναι απλώς ε, τροπολογίες διαγραφής να τις ψηφίσουμε μπλοκ. Γίνεται. Θα προτείνω κάτι εντό ολίγου. Θα σας προτείνω ακριβώς αυτό, διότι όλες οι ε, ψηφοφορίες συμπίπτουν. Η 58 εγκρίνεται. 59 υπέρ. Ah, συγγνώμη, ήμασταν στην 56 εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές αποσύρεται. Ε, ε απορρίπτεται, συγγνώμη. 58 του κυρίου Σαρβαμά με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ή 60. Επειδή το αποτέλεσμα είναι ταυτόσιμο στις ε, τροπολογίες διαγραφές των διαφόρων παραγράφων ή τμήματων των παραγράφων, προτείνω από εδώ και πέρα οι τροπολογίες της κυρίας Μοντέλ να θεωρήσουμε ότι απορρίπτονται. Συμφωνούμε? Ωραία. Η 61 αποσύρεται. Συγγνώμη, 61 απορρίπτεται, 62 απορρίπτεται, 63 επίσης, 64 επίσης, 65, η 66 απορρίπτεται. Για την τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 69 απορρίπτεται, 70 απορρίπτεται, 71 απορρίπτεται, η 72 αποσύρθηκε, 73 απορρίπτεται, 74 αποσύρθηκε, 75 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 76 απορρίπτεται. 77 καταπίπτει. 78 απορρίπτεται, 79 απορρίπτεται, 80 απορρίπτεται, 81, 82, 83 απορρίπτονται, 84 κατέπεσε. Η ετρία e εγκρίθηκε, επομένως καταπίπτει. 85 απορρίπτεται, 86 απορρίπτεται, 87. Ψηφίζεται. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88 ε, απορρίπτεται, 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 90 Απορρίπτεται 91. Απορρίπτεται 92, 93, 94, 95, 96, 97. Απορρίπτονται 98. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 99, 100, 101, 102, 103, απορρίπτονται 104. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 105, 106, 107, 108 απορρίπτονται, 109 απορρίπτεται, 10, 111 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 112 απορρίπτεται, 113, 114, 115, 116, 117, 118 επίσης, τροπολογία 4 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται.

αποχές απορρίπτεται 132, 133 καταπίπτουν 134, 135 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 137 απορρίπτεται 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 160, 151, 100 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οι άλλες ε, έχουν απορριφθεί. 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 172 απορρίπτεται, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183. Πάμε στην 192. Συγγνώμη, Πάμε στην 192 υπέρ, κατά, αποχές, α, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 5 απευθεία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 203 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 218 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 225 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 127 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 229 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 231 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 233 υπέρ, κατά, πανομοιότυποι, απορρίπτονται, 242 υπέρ, κατά αποχές καταπίπτει 245 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 248 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 256 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 265 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία παριθμών 7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη. 271 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 274 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 278 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 284 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 285 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 288 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 292 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 304 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περνάμε σε αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 18 ψήφοι κατά, 14 υπέρ. Ήταν η 8. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Όχι. Λάθος, συγγνώμη, όχι τη 13. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 απορρίπτεται, 23 επίσης, 24. Τροπολογία 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα στο σύνολο του κειμένου. Πρέπει να γίνει μια διόρθωση. ψηφίσαμε την 3 και η 3 σήμαινε ότι πρέπει να ψηφιστεί και η 75 και επομένως πρέπει να διορθωθεί η ψηφοφορία για το 75 και θα ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου λοιπόν ως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 30 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά. Συγχαρητήρια στο συντάκτη της γνωμοδότης, τον κύριο Γκάιερ. Και πάμε τώρα να ψηφίσουμε για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη Επαγγελματικής Κατάρτισης, το ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Η κυρία Μοντέλ και πάλι έχει καταθέσει πάρα πολλές τροπολογίες. Στόχος είναι η κατάργηση του οργανισμού και η πρώτη τροπολογία αφορά τον τίτλο. Επομένω, εάν καταψηφίσετε την τροπολογία τη κυρία Μοντέλ, θα θεωρήσουμε ότι όλε οι τροπολογίε τη κυρία Μοντέλ που ε, αφορούν ε, τι παραγράφου μπορεί να θεωρήσουμε ότι απορρίπτονται από την Επιτροπή. Ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και αυτό σημαίνει ότι θα μεταφραστεί η ψήφος στην άποψή σας. Ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας της κυρίας Μοντέλ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται λοιπόν, επομένω όλε ε, οι τροπολογίε ε, τη κυρία Μοντέλ ε, απορρίπτονται και για τα άρθρα και για τι παραγράφου κτλ. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 43. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 3 αποσύρεται. Η 50 καταπίπτει. 51. Με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67. Άρα τι έγινε με την 4. Εγκρίθηκε. Άρα η 67 καταπίπτει. Καθώς και 68. Περνάμε στην 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. «149. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 150 όχι καταπίπτει. 153 υπέρ. 150 μάλλον. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 163 του κυρίου Σαρβαμά. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 209. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 10. Περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και για το σύνολο του κειμένου. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Όχι, όχι, όχι. Α, ζητώ συγγνώμη. Τροπολογία 11. Είναι επί της διατύπωσης 12 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 13 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 14 καταπίπτει, 15 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 16 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά εγκρίνεται. 20 υπέρ α καταπίπτει. 19 καταπίπτει επίσης. 22 υπέρ καταπληκτική 22, 24 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Για το σύνολο του κειμένου ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται. Πέρας. με 30 ψήφους υπέρ, 2 κατά, συγχαρητήρια. Περνάμε τώρα... Α, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, εν συντομία, να σχολιάσω κάτι. Ε, υπάρχει ε, ακόμα ένα ζήτημα με τις... Υπήρχαν μόνο πολλές τροπολογίες που μας δημιούργησαν πρόβλημα, αλλά χάρη ε, στις ε, τροπολογίες της κυρίας Μοντέλ βελτιώσαμε και τα γαλλικά μας. Θα ήθελα να υπάρχει ένα πρόβλημα με την ε, διερμηνία. <laughs> Και τα έλεγα τόσο ωραία. Ήθελα να πω μόνο αυτό, ότι συνάδελφοι, ήταν πολύ καλέ οι τροπολογίε ε, τη κυρίας Μοντέλ γιατί με βοήθησαν ε, να βελτιώσω τα, τα γαλλικά μου, διορθώνει ο μιλητή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για να το κάνω αυτό πρέπει να μάθω τα νούμερα. Ε, ακόμα μου δημιουργεί πρόβλημα το 80 που είναι λίγο περίπλοκο στα γαλλικά. Κάποιο όμω πρέπει να εξηγήσει στην κυρία Μοντέλ ότι όλε αυτέ οι τροπολογίε είναι ανόητε. Και το να προτείνει να διαγράφεται κάθε παράγραφος, ποιος είναι ο σκοπός. Και σας παρακαλώ να μιλήσετε με την ε, κυρία Μοντέλ για αυτές τις τροπολογίες για να σταματήσει αυτό το παιχνίδι, γιατί πραγματικά είναι απαράδεκτο. Εδώ εξοδεύουμε και χάνουμε χρόνο για αυτή την ανοησία. και πραγματικά προτείνω κάποιος από τη γραμματεία να πάει στην κυρία Μοντέλ και να της πει εντάξει καλά έκανε και τα έβαλε όλα αυτά τα νούμερα στα γαλλικά αλλά πρέπει να σταματήσει εδώ. Montel. Ε, ναι, δεν είναι εδώ η κυρία Μοντέλ. Κάποιες φορές την βλέπουμε. Παρακαλώ κύριε Μακά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ άκουσα τα όσα είπε ο συνάδελφο και τα αντιλαμβάνομαι. Αλλά αν συζητούμε γι' αυτό θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη μας ε, όλες τις τροπολογίες. Ε, δηλαδή πρόκειται για ζήτημα στατιστικών στοιχείων αν θέλετε. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε μια άθρηση όλων των τροπολογιών ε, αναβουλευτή. Εν πάση περιπτώσει για την ε, κυρία Μοντέλη, η οποία υποβάλλει σε αυτές τις τροπολογίες, έχει νόημα. Ε, εντάξει, ορισμένες φορές μπορούν οι δείκτες επιδόσεων να ε, μας ε, οθήσουν στα εργαλεία ε, βελτιστοποίησης και αυτό μπορεί να, πραγματικά να αποβεί γελίο. Όλα αυτά έχουν ένα κόστος βέβαια. Για το πνεύμα των τροπολογιών, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Εγώ προέρχομαι από την ίδια πολιτική ομάδα ε, και ακόμα και εγώ ενοχλούμαι από αυτές τις ε, από αυτή τη των τροπολογιών και δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. δεν ξέρω και ποια είναι η σχέση της ε, κυρίας αυτής με το Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά σε κάθε περίπτωση πραγματικά και εγώ πιστεύω ότι στην πράξη δεν θα πρέπει να επαναληφθεί αυτό στο μέλλον, γιατί δεν δίνει και καλή εικόνα και για μας. Ευχαριστώ. Ήθελα και εγώ πολύ σύντομα να πω ότι ε, υπάρχει ελπίδα ότι σε δύο μήνε θα επιληθεί από μόνο του το ζήτημα και από εκεί και μετά υπάρχει και αυτό που είπε ο συνάδελφο Σιμάνκα. Δηλαδή, είναι δύσκολο να παριθμούμε μόνο ε, εγκεκριμένε, αν θέλετε, τροπολογίε. Ε, ίσως θα μπορούσε Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών να τοποθετηθεί επ, αυτού του ζητήματος ε, δηλαδή ε, σε ό,τι αφορά τις συνολικές τοποθετήσεις και την διάθεσή τους στις διάφορες rating agencies. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να δώσουμε μια, ένα σχετικό έναυσμα εδώ ως Επιτροπή του Προπολογισμού και πολύ σωστά είπε και ο Πρόεδρος ότι ε, η μετάφραση των τροπολογιών που προτείνουν διαγραφές είναι πολύ εύκολη. Αντιθέτως όμως όταν έχουμε τροπολογίες οι οποίες ε, περιλαμβάνουν διάφορα κείμενα copy-paste πραγματικά εκεί ε, το κόστος φτάνει στις χιλιάδες ευρώ και εκεί τίθεται ένα ζήτημα του κατά πόσο έχει νόημα κάτι τέτοιο ή όχι. Ναι, ήθελα μόνο να επισημάνω στους αδέλφους ότι όλοι μας πρέπει να πληρώσουμε το τίμημα για να παραμείνει δημοκρατική ε, η Γαλλία. Καλύτερα λοιπόν να ψηφίσουμε εδώ τις τροπολογίες παρά να την έχουμε στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Alors, vrai que... Πράγματι, πρόκειται για να αναφέρω το δικαίωμα το, αυτό της υποβολής ε, και κατάθεσης τροπολογιών όμως, όπως ε, και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα, θα πρέπει να προχωρούμε σε καταχρήσεις. Πρέπει να γίνεται με μέτρο η αξιοποίησή του. Η γραμματεία λοιπόν ε, προσέγγισε την κυρία Μοντέλ και ήθελε η Επιτροπή Προπολογισμού να κατανοήσει το το κόστος που ενέχουν αυτοί οι οργανισμοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνω λοιπόν την επόμενη φορά να τη στείλουμε ένα, ε, να μας στείλει ένα μικρό μήνυμα και να μας πει ότι κατανοούμε αυτό το κόστος, αλλά να πούμε και εμείς ότι το κόστος ε, της μετάφρασης ε, των τροπολογιών είναι ακόμα μεγαλύτερο ίσως. Και ότι όλα αυτά παίρνουν χρόνο και ενέργεια και θυμίζει το filibustering που υπάρχει στην Αμερική και κατανοείται πόσο μας δυσκολεύουν τα πράγματα. Τώρα ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ευχαριστώ τον συνάδελφο για την ε, επισήμανση που έκανε. Αν η κυρία Μοντέλ ερχόταν πιο συχνά στις επιτροπές θα μπορούσε να μας μιλήσει κιόλας γι' αυτό. Ωραία πάντως που έτσι ξεσπαθώσαμε λίγο. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο θέμα, Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Βίωση και Εργασία, Eurofound. Και εδώ κυρία Μοντέλ έχει πολλές. Κατανοήσαμε την, οδηγία, την, ε, ε, την ίδια μέθοδο θα ακολουθήσουμε και τώρα. Αν μπλοκ θα ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες διαγραφής για τις ε, παραγράφους, τα άρθρα και τις παραγράφους και τα τμήματα παραγράφων. Θα ψηφίσουμε για την 21 λοιπόν και ανάλογα με τη στάση θα θεωρήσουμε ότι ακολουθεί την ίδια στάση και για τις υπόλοιπες τροπολογίες τη κυρίας Μοντέλ. Γνωρίζουμε ότι η 206 ε, είναι απαράδεκτη. Μη παραδεκτή τέλος πάντων. Για την 21, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, Επομένω, ε, απορρίπτονται όλε οι τροπολογίε διαγραφή τη κυρία Μοντέλ. Μάλιστα, περνάμε στην 34 του κυρίου Σαρβαμά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι δύο αποσύρεται. 37. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36 αποσύρεται. Η 37 καταπίπτει, καθώς και 40, 41. Υπέρ. Α, ναι, καταπίπτει. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 53 καταπίπτει εφόσον εγκρίθηκε η 3. me t il Amendement numéro 4. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παίρνουμε τώρα, τώρα στις αιτρολογικές σκέψεις. Οι 8 και 9 καταπίπτουν. 10. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11, 12, 13 καταπίπτουν. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Καταπίπτουν 14 και 15. 17. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίσουμε επί το συνόλου του κειμένου, όσο έχει τροποποιηθεί, άρχεται ψηφορία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, επιθυμίζω. Πέρας. Εγκρίνεται με 30 ψήφους υπέρ, 2 κατά. Σε στον εισηγητή Γιάννη Σκάιερ. Ε, για το 14 δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν τήσεις μεταφοράς, οπότε δεν υπάρχει νόημα, ούτε για το 15, ούτε για το 16 της κυρίας Χολμάιερ. Επομένω κλείνει εδώ η ψηφοφορία. Εάν δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, θα σταματήσουμε εδώ. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 4. Με οποιονδήποτε θέλει να προεδρεύσει. Εμένα θα με συγχωρήσετε, αλλά πρέπει να φύγω. Θα πάω στο Παρίσι και θα επιστρέψω το πρωί. Τα ξαναλέμε στις 4 μάλλον. Εσείς μάλλον θα συνεχίσετε.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Ο πρόεδρος μας, ο κύριος Αρτουή, χρειάστηκε να αποχωρήσει και μεταξύ των αντιπροέδρων ε, είχα εγώ την τιμή να προεδρεύσω σε αυτή τη συνεδρίαση ε, εκτάκτος. Ε, ξεκινούμε λοιπόν αυτή τη δημόσια ακρόαση για την χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων και τη σύνδεσή τους με άλλα επενδυτικά ταμεία. Ο λόγος ε, και πάλι καταρχάς ε, στον εισηγητή, τον κύριο Φερνάντες. Κύριε Φερνάντες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι τιμή να σας έχω ε, Πρόεδρο. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Νομίζω πως ε, όλοι μας γνωρίζουμε ότι τα διαφορετικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής ε, και το Ταμείο για την Περιφερειακή Αναδούση στο Ταμείο για την Αλληλεία είναι ταμεία πάρα πολύ σημαντικά τα οποία θα πρέπει να ε, συμπεριλαμβάνονται στις εταιρικέ σχέσεις και στα κατάλληλα χρηματοδοτικά ε, μέσα. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορούμε ε, να υποτιμήσουμε την σημασία κανένας από αυτά τα επιμέρους ταμεία. Και αυτή είναι η σημαντική πρόκληση για εμάς. Δηλαδή να ακούσουμε σήμερα από τους εμπειρογνώμονες εάν πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα και να ακούσουμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερες συνέργειες, μια υψηλότερη αξιοποίηση των κοντιλίων αυτών των ε, ταμείων, πώς μπορούμε δηλαδή να αντλήσουμε αν θέλετε περισσότερο αντίκτυπο μέσω μιας καλύτερης εκτέλεσης αυτών των διαφθορτικών ε, ταμείων. Με ποιον τρόπο δηλαδή μπορούμε στο μέλλον να προχωρήσουμε στην καλύτερη αξιοποίηση χωρίς να υποβαθμίσουμε ούτε ε, τα χρηματοκροτικά εργαλεία, ούτε τα ε, επενδυτικά ε, και τη ταμεία. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνεχής θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη σημασία που έχουν και σήμερα. Ε, και ε, θα πρέπει να πω ότι ε, ορισμένες φορές έχω αντιμετωπίσει δυσκολίες στο να εξηγήσω ε, Στου συναδέλφου μου για παράδειγμα στην Πορτογαλία ω προ το τι συμβαίνει σε σχέση με τα διευθυντικά ταμεία και ότι δεν δηλαδή βρίσκονται παρόντα στη δική μα χώρα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στις υποδομές. Ε, δηλαδή υπάρχει μεγάλη χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά το επίπεδο των επιχειρήσεων τη ενέργεια και αλλού, αλλά δεν υπάρχουν επενδύσει στι υποδομέ. Άρα λοιπόν ε, ακριβώς σε αυτό το επίπεδο χρειαζόμαστε τα συμπληρωματικά χρηματοδοτικά εργαλεία που θα πρέπει να αξιοποιούμε. μια ακόμα ε, σημαντική ερώτηση που θα ήθελα να θέσω στους εμπειρογνώμονες, ήδη άρχισα δηλαδή να θέτω ερωτήματα, είναι ποια είναι η επικοινωνία, ποιος είναι ο συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Για παράδειγμα, ε, τι ε, μπορεί να γίνει σε επίπεδο σύνδεσης του ΕΦΣΙ, του Ταμείου Στατηγικών Επενδύσεων, στο επίπεδο του στο επίπεδο άλλων ε, ε, ε, σε σχέση με το συντονισμό τους με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να αποφύγουμε την επικάλυψη των εργασιών. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι έχουμε την καλύτερη κοινή αντιχρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, η Ευρώπη χρήζει περαιτέρω επενδύσεων. Αν δούμε δηλαδή τον αντίκτυπο του Ταμείου Στατικών Επενδύσεων θα δούμε ότι ήδη έχουμε πολύ ε, θετικές επιπτώσεις και σε επίπεδο επενδύσεων γενικά και στο επίπεδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αναμένουμε να υπάρξει και ακόμα ε, πιο σημαντικός αντίκτυπος και πιο ορατός αν θέλετε, πιο προβλημένος. Γιατί συχνά ούτε επιχειρήσεις ούτε ο πληθυσμός γνωρίζουν ακριβώ το τι έχει γίνει, ποια υποστήριξη έχει δοθεί. Για παράδειγμα, ήδη 400.000 επιχειρήσει έχουν επωφεληθεί από το ΕΦΣ και γενικά την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα. Από εκεί και μετά, οι επιμέρους πλατφόρμες που υπάρχουν, πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Πώς μπορούμε ταυτόχρονα να προωθήσουμε περισσότερο τις εταιρικέ διασυνοριακές σχέσεις, γιατί τέτοιου είδους διασυνοριακά στοιχεία είναι ε, ε, εξαιρετικά απαραίτητα ε, ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στον τομέα τη ενέργεια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε καλύτερα να αξιοποιήσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα διαθωτικά ταμεία ε, προ αυτό το σκοπό. Και από εκεί και μετά βέβαια μια σημαντική προτεραιότητα για μέσα είναι να αποφύγουμε την περιφερειακή συγκέντρωση. Δηλαδή θα πρέπει το ΕΦΣΥ να προσαρμοστεί στις προτεραιότητες αν θέλετε της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει δηλαδή να υποστηρίζουμε την συμπληρωματικότητα προφανώς, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να λαμβάνεται υπόψη και η ρεαλιστική διάσταση, αν θέλετε, ενός ε, έργου. Δηλαδή δεν είναι η ίδια η σημασία ε, ενός έργου στα διαφορετικά κράτη-μέλη και μάλιστα σε μέρους περιοχές ενδεχομένως του κάθε κράτους μέρους. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο αντίκτυπος να λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με τις επιμέρους κατά τόπου ιδιαιτερότητες προκειμένου να ε, εφαρμόζεται για παράδειγμα ένα κίνητρο ή μια συγκεκριμένη εξαίρεση στο πλαίσιο ενό κανονισμού προκειμένου ακριβώς να λαμβάνονται υπόψη αυτές οι ιδιαιτερότητες και να αξιοποιείται λοιπόν στο πλαίσιο της ε, πολιτικής ε, συνοχής καλύτερα το τι μπορεί να μας δώσει το ΕΦΣΥ. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου, όσο χρειάζεστε. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Θα συνεχίσω στα πορτογαλικά. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της πραγματικότητας. Όπως είπα, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την ε, πραγματικότητα, τι ισχύει δηλαδή σε επίπεδο περιφερειακής ιδιαιτερότητας. Κάτι το οποίο δεν έχει ληφθεί ακόμα δεόντως υπόψη κατά την άποψή μου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την προεπιλογή ε, των ε, έργων. Ε, μία προτεραιότητα που σχετίζεται με αυτό είναι το πώς μπορούμε να συμπεριλαμβάνουμε πάντα στις επενδύσεις τα έργα εκείνα τα οποία μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Γιατί η Τράπεζα Επενδύσεων προβλέπει την χρηματοδότηση μέσω του ΕΦΣ έργων ε, τα οποία ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία έχουν πολύ σημαντικό αντίκτυπο που δεν πληρούν αυτό το κριτήριο και θα πρέπει λοιπόν να ε, διασφαλιστεί η ε, συγχρηματοδότησή τους μέσω του ΕΦΣΥ. Αυτές είναι λοιπόν οι αμφιβολίες μου. Αυτά είναι τα ενάβασματα αν θέλετε που δίνω προς σκέψη ως προς τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Τη δουλειά δηλαδή που έχει γίνει, χρήσιμη πραγματικά δουλειά και επιτρέψτε να πω και κάτι τελευταίο. Αυτό το earmarking στο οποίο εγώ αντιτίθεμαι αν θέλετε, το οποίο εφαρμόζεται και εδώ και μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές, σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν και τέτοιου είδους οριζόντιες ε, διαστάσει που θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μα. Άρα λοιπόν υπάρχουν μία σειρά από συστάσει τι οποίε θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε για το εύση δεύτερη γενιά, το εύση 2 δηλαδή. οι επενδύσεις εκείνες οι οποίες είναι χρήσιμες ε, για την ε, ε, κοινωνία και την οικονομία, δηλαδή προωθούν την οικονομική ανάπτυξη και είναι ταυτόχρονα και βιώσιμα, θα πρέπει να λαμβάνουν την κατάλληλη υποστήριξη. Εκτός και αν βέβαια ε, υπονομευθούν, αν θέλετε, από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν και από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ευχαριστώ λοιπόν ε, για την διοργάνωση της σημερινής ακρόσης και για την παρουσία των εμπειρογνωμών σήμερα Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φερνάντες για αυτή την εισαγωγή, η οποία ήταν και υπομορφή ερώτησης, αλλά ταυτόχρονα και έκκλησης, διότι αν κατάλαβα καλά, η ερώτηση περιέλαμβανε και μία έκκληση. Να περάσουμε τώρα στους ομιλητές μας. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να δώσουν μια απάντηση συνολικά στην ε, ερώτηση που έθεσε ο εισηγητής. Ο Ερικ Φον Πρέσκα έχει πρώτο το λόγο από τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Προφανώς δεν είμαι σε θέση να απαντήσω όλες αυτές τις ερωτήσεις που ετέθησαν από τον εισηγητή. Αυτό που προτείνω λοιπόν είναι να ε, κάνω μια σύντομη αναφορά ε, στα της εφαρμογής ε, των διαρθρωτικών ταμείων τώρα κατόπιν να δούμε εντάχει και τα διδάγματα τα οποία αντιλήσαμε, τι πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να αλλάξει στο μέλλον και στο τέλος θα πρέπει να πω δύο λόγια και για τις συνέργειες και τις συμπληρωματικότητες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και φυσικά ε, και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, το ΕΦΣΥ που νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει περισσότερο. Ε, να σας πω λίγο σύντομα πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ δύο μορφών προγραμμάτων. Τα πρώτα είναι προγράμματα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013 όπου είμαστε στη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Τα κράτη-μέλη πριν από κάποιες εβδομάδες μάλιστα υπέβαλαν τα τελευταία αιτήματα πληρωμής και τα έγγραφα ε, για την καθάριση και θα δείτε ότι τα περισσότερα, αν όχι τα ε, όλα τα κράτη-μέλη, είναι στο 95% ποσοστού εκτέλεσης. Στα αριστερά έχετε την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα ε, έχερε ειδικών κανόνων λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης και στα δεξιά έχετε την Κροατία, η οποία είναι σε χαμηλότερο βαθμό από τους υπολείπους, γιατί η Κροατία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013. Επομένως έχουν λίγο περισσότερο χρόνο για να ταπανίσουν τα κονδύλια. Αυτό είναι ε, μια επιτυχημένη ιστορία, ιδιαίτερα αν δείτε και τα στοιχεία εφαρμογής όσον αφορά τα επιτεύγματα διότι όταν λαμβάνουμε τις πληροφορίες από τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να μας υποβάλουν και εκθέσεις για τα φυσικά προσκόμματα και τα επιτεύγματά τους. Και από αυτό που γνωρίζουμε από τα προγράμματα μέχρι το 2013 είναι ότι πάνω, δημιουργήθηκαν πάνω από 1,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και επίσης ένας άλλος δείκτης που είναι σημαντικός πάνω από 50 εκατομμύρια επιπλέον ε, νοικοκυριά έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικό δίκτυο λόγω των επενδύσεων που είχαμε από τα διαφορετικά ταμεία. Για το πρόγραμμα τώρα 2014-2020 ε, τα στοιχεία δεν είναι ακόμα τόσο θετικά δυστυχώς, διότι αν δείτε το ποσοστό οικονομικής εκτέλεσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως δαπάνες από τον προϋπολογισμό και φαντάζομαι ότι η Επιτροπή σας τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό, το 2016 είχαμε απόδοση κάτω το αναμενόμενο. Δεν μπορέσαμε να απορροφήσουμε όλο το διαθέσιμο προπολογισμό. Το θετικό βέβαια είναι ότι αν δούμε την κατάσταση επιτόπου, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ε, μια πολύ μεγάλη επιτάχυνση. Επιτάχυνση όσον αφορά τα προγράμματα τα οποία επελέγησαν, ε, και όπως γνωρίζετε πάντα χρειάζεται λίγος χρόνος μέχρι να υποβάλουν τις τελικές αιτήσει πληρωμής ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, οι υπεύθυνοι των έργων, αλλά θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ προγραμμάτων έχουν προεπιλεγεί και είναι στη διαδικασία της υλοποίησης και θα δείτε επίσης ότι ε, στο διάγραμμα αυτό ότι χοντρικά αυτό αφορά το 1 τρίτο της κατανομής των ποσών αλλά θα δείτε ότι υπάρχουν και μεγάλες ε, διαβαθμίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Κάποια είναι πολύ προχωρημένα όσον αφορά την επιλογή των προγραμμάτων και κάποια άλλα υστερούν. Επομένως, ε, σίγουρα υπάρχει δουλειά να γίνει για να μπορέσουν να προλάβουν τους υπολείπους, ώστε να διασφαλίσουμε και ότι θα ε, επιταχύνουμε την ε, υλοποίηση των προγραμμάτων. Για ποιο λόγο υπάρχει καθυστέρηση. Ένας από τους βασικούς λόγους, και μάλιστα αυτό αποτελεί ίσως και ένα δίδαγμα για το μέλλον, ε, είναι ότι καθυστέρησε η έγκριση του νομοθετικού πλαισίου, η οποία έγινε τα μέσα Δεκεμβρίου του 2013, που σημαίνει ότι είχαμε και μία καθυστέρηση στην έναρξη των νέων προγραμμάτων, Άρα αυτό σημαίνει ότι την επόμενη φορά, δηλαδή για το μέλλον μετά το 2020, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μην έχουμε τέτοιες καθυστερήσεις. Κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας ε, είναι το γεγονός ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο επικεντρώνεται πάρα πολύ στην ποιότητα, πολύ περισσότερο στην ποιότητα από ότι το προηγούμενο. Αυτό βεβαίω σημαίνει ότι πολλοί από τους διαχειριστές των προγραμμάτων θα πρέπει να κάνουν επιπλέον δουλειά πριν ε, να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση πληρωμής ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σημαίνει με τη σειρά του ότι υπάρχει ε, ένα χρονικό κενό μέχρι να ξεκινήσουν να υποβάλλονται οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, αποζημίωση των δαπανών. Και τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, το οποίο θα πρέπει να έχετε κατά νου, υπάρχουν αρκετές νομοθετικές αλλαγές οι οποίες ε, δεν μας χαροποιούν ιδιαίτερους. Για παράδειγμα, ο αυτόματος κανονισμός αποδέσμευσης από τα δύο πήγε στα τρία χρόνια, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κίνητρα για τα κράτη-μέλη και τις αρχές να εφαρμόσουν ε, ταχύτατα ε, και να προχωρήσουν τις επενδύσεις. Και κάτι τελευταίο, ε, υπάρχει και έλλειψη διοικητικών δυνατοτήτων στα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει δηλαδή ε, επάρκεια προγραμμάτων ε, και ε, έλλειψη και διοικήσεων που να είναι σε θέση να προχωρήσουν πολύ γρήγορα. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι για μας η προτεραιότητα το 2017 είναι να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και τους διαχειριστές προγραμμάτων όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση ώστε να μπορέσουν να επιταχύνουν. Γίνεται λοιπόν στενή παρακολούθηση από πλευρά μας και επίσης τους βοηθούμε για τη δημιουργία διοικητικών ικανοτήτων με συγκεκριμένα μέτρα να βοηθήσουμε αυτές τις διοικήσεις και να βοηθήσουμε και τις προβλέψεις των πληρωμών. Γιατί τελικά αυτά τα οποία υποβάλλουμε στο Κοινοβούλιο εξαρτάται από αυτά τα οποία λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη όσον αφορά τον προπολογισμό που απαιτείται για την άντληση των απαραίτητων πόρων. Και τέλος, κάτι το οποίο έχουμε βάλει και στο διαδίκτυο, ε, έχουμε μία ανοιχτή πλατφόρμα δεδομένων, στην οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε ε, σε πραγματικό χρόνο την εφαρμογή επιτόπου. Η ιδέα είναι να υπάρχουν κάποια ορόσημα και κάποια ε, εξέταση μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μεγάλη διαφάνεια στο θέμα της εφαρμογής. Περνάω τώρα στο επόμενο σημείο. Ποιες είναι οι ιδέες μας για το μέλλον στον τομέα αυτό. Και όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις ξεκίνησε μια διαδικασία περισυλλογής για το μέλλον της Ευρώπης και το επόμενο βήμα είναι ένα έγγραφο περισυλλογής για την χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο νομίζω θα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δεύτερο 15 ε, του Ιουνίου, όπου θα παρουσιάσουμε κάποια ανάλυση για το μέλλον, αλλά βεβαίως δεν περιμένουμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο για το 2020 και μετά θα παρουσιαστεί πριν από το 2018. Ακόμα λοιπόν απέχουμε από ε, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ελπίζουμε ότι θα λάβουμε και αρκετά στοιχεία από εσά και πολλές πληροφορίες και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν ε, αυτό δεδομένου ότι είστε και συνομοθέτης για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την επόμενη ε, δέσμη μέτρων σε νομοθετικό επίπεδο. Κάτι ακόμα το οποίο είναι σαφές είναι η απλοποίηση του συστήματος διαχείρισης, ε, διότι πιστεύουμε ότι σε κάποιους τομείς έχουμε υπερβεί λίγο τα όρια και ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή και είναι και σημαντικό να απλουστεύσουμε λίγο την νομοθεσία και να μειώσουμε το άχθος για τους διαχειριστές των προγραμμάτων και να υπάρχει και μεγαλύτερη ευελιξία. Πρόκειται σαφώς ε, για κάτι που μας απασχολεί. Πέραν αυτού το θέμα είναι και μέχρι ποιο βαθμό είναι λογικό να αλλάξουμε το σύστημα διαχείρισης, διότι Υπάρχουν κάποιες επικρίσεις σε κάποιες ε, περιοχές για την κοινή ε, τη συνδιαχείριση, για το πώς εφαρμόζονται, αλλά το να αλλάξουμε τρόπο διαχείρισης σημαίνει ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές αλλαγές, ίσως και μεγάλη αβεβαιότητα και καθυστερήσεις. Άρα το ερώτημα όντως είναι μήπως καλύτερα θα ήταν αντί να μεταρρυθμίσουμε εκ νέου το σύστημα, να πούμε ότι η καλύτερη μεταρρύθμιση είναι να μην αλλάξουμε τίποτα, ώστε τα κράτη-μέλη και οι αρχές τους, τώρα που γνωρίζουν τους κανόνες, να είναι σε θέση απλώς να ε, προχωρήσουν και να μετακυλήσουν το σύστημα διαχείρισης και να μην τα φέρουμε όλα πάνω κάτω από την αρχή. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά φυσικά και μαζί σας και με άλλους ενδιαφερομένους. Και εδώ έρχομαι στο τελευταίο σημείο, συνέργειες με άλλα μέσα. Το πρώτο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω εδώ είναι ότι ο συνδυασμός με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ, ήδη ε, επιτρέπεται. Αλλά επειδή ο κανονισμός για τα διορθωτικά ταμεία εγκρίθηκε πριν από τη δημιουργία του ΕΦΣΥ, υπάρχουν αρκετοί συνδυασμοί οι οποίοι δεν επιτρέπονται αυτή τη στιγμή ε, βάσει των νόσων ισχύων. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε προτείνει και αυτό το οποίο ε, έχετε ίσως συζητήσει ήδη, η λεγόμενη πρόταση Omnibus. Η πρόταση Omnibus περιλαμβάνει επιπλέον προϋποθέσεις για να έχουμε τα επιπλέον κονδύλια, γιατί ένα από τα βασικά θέματα τα οποία διαπιστώνουμε με το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι ότι υπάρχουν κάποιε περιοχέ και κάποια μέρη τη Ευρώπη όπου είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί, διότι είναι πολύ μεγάλο ο κίνδυνο. Και το σκεπτικό με τι αλλαγέ που προτείνουμε είναι τα διαρθρωτικά ταμεία και το ΕΦΣΥ να συνδυαστούν και να μπορούν τα διαρθρωτικά ταμεία να αναλάβουν ε, αυτό το λεγόμενο first loss piece, δηλαδή να αναλαμβάνουν τον κίνδυνο για να μπορούν να χρηματοδοτούνται προγράμματα τα οποία σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν από το Ταμείο Στρατηγών Επενδύσεων. Έχετε κάποια ερώτηση? Όχι, συγγνώμη. Τρεις φράσεις ακόμα. Μας εξέπλησε λίγο η αρνητική στάση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το συγκεκριμένο. Διότι και στο Συμβούλιο αλλά και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η αρχική αντίδραση ήταν μάλλον χλιαρή θα έλεγα διότι από ό,τι καταλάβαμε, θεωρήθηκε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ευνοεί πολύ την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ε, εις βάρος των διαθροτικών ταμείων. Μετά από πολλές συζητήσεις και εξηγήσει, βέβαια, ε, διαπιστώνουμε τώρα ότι και το Συμβούλιο αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αντιληφθεί ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σωστή και θα την υποστηρίξουν και τα δύο θεσμικά όργανα. Και για μας αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι θέλουμε ε, να μπορέσουμε να έχουν αποτελεσματικούς νέους συνδυασμούς και το συντομότερο δυνατόν. Γι' αυτό ακριβώς και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία πριν από το τέλος του έτους. Επαναλαμβάνω, για μας ε, δεν τίθεται θέμα εύσης βάρος των διαρθρωτικών ταμείων. Θέλουμε να συνδυάσουμε δύο χρηματοδοτικά μέσα σε καιρούς που είναι δύσκολα γιατί υπάρχει σπάνιδη, σπάνιδα ε, ε, δημοσίων πόρων και υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες δεν θα είχαν πρόσβαση στο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ε, γιατί κάποιοι ενδότες επενδυτές μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι πολύ επικίνδυνη η επένδυση και επομένως θα γίνουν αυτές οι αλλαγές όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Βονμπρέσκα, επιτρέψτε μου να προσθέσω εδώ μια προσωπική σκέψη και μόνο, ε, που δεν έχει καμία σχέση με την ουσία. Νομίζω πρέπει να αλλάξω γυαλιά μάλλον. Γιατί δεν βλέπω καν μέχρι την ε, οθόνη. Ε, ίσως ε, βέβαια και εσείς θα μπορούσατε να μας ε, δείξετε πιο ευανάγνωστους πίνακες. Ο κύριος Φερνάντες και στην αρχική του παρέμβαση περιμένει κάποια στοιχεία που θα απαντήσουν στα δικά του ερωτήματα. Εγώ δεν τα είδα προσωπικά, αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ντέιβιτ Σκόρνια. Συγγνώμη αν ε, δεν προφέρω στο το όνομά σα. Είναι διευθυντή αρμόδιο για ζητήματα εταιρικών σχέσεων, εξολογήσεων και στρατηγικών στο ε, Υπουργείο Περιφερειακή ε, Ανάπτυξη τη Τσεχία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ladies and gentlemen. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σεγητά, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω την ευγνωμοσύνη μα που μα επιτρέπετε να παρουσιάσουμε τη δική μα προοπτική σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή και να σα ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και τα ερωτήματα που εγείρατε. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να επισημάνουμε τον ρόλο της πολιτικής συνοχής πριν ε, σας παρουσιάσω πώς έχει κατάσταση σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή της ε, και την προοπτική για το μέλλον. Θεωρούμε ότι καλύπτει αρχικά την δέσμευση της ε, εκτέλεσης ενός ευρωπαϊκού προπολογισμού με βάση τα αποτελέσματα. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά μέσα ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Θεωρούμε ότι η πολιτική συνοχής λοιπόν είναι πολύ σημαντικός άξονας ε, ανάπτυξης. Έχει αποδείξει ε, τον ρόλο κλειδί που διαδραματίζει ακόμα και σε μια περίοδο ε, κρίσης τα τελευταία χρόνια. πλέον ε, είναι πιο προβλημένη και ορατή η πολιτική ε, στις επιμέρους χώρες και συμβάλλει στην ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Have a little technical trouble with... Uh, yeah, okay, good, good. Uh, we think the, uh, uh we would like to uh, uh, point your attention to... Θα θέλαμε να ευχηθήσουμε την προσοχή σας σε πραγματικές ε, αλλαγές που έχουμε και στην Τσεχία, γιατί το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα. γιατί θεωρούμε ότι έτσι ε, εξυπηρετούμε και τον βασικό σκοπό της πολιτικής συνοχής, όμως ταυτόχρονα η πολιτική συνοχής βελτιώνει ε, και τη στρατηγική διοίκηση, τον σχεδιασμό οριζόντων και των εταιρικών σχέσεων. Και ίσως αυτό δεν είναι ο αρχικός ίσως ε, στόχος που είχαμε θέσει, όμως βλέπουμε ότι επιτυγχάνονται. Θα σας δώσω και ορισμένα στοιχεία τώρα. Στην πρώτη εικόνα βλέπετε την πραγματική σύγκληση των ε, περιφερειών ε, της στοιχείας βάσει του περιφερειακού ΑΕΠ, κατά ΑΕΠ, από το 2004 μέχρι το 2014. Βλέπετε είναι μια σημαντική σύγκληση και είχαμε 4% παραπάνω ε, με το 2015, 3% κάτω ενεργεία. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 34% όλων ε, των κεφαλακών επενδύσεων της κυβέρνησης προκύπτουν από ε, τα διαφορετικά και επενδυτικά ταμεία. Αυτό λοιπόν αυξάνει τη σύγκληση μεταξύ των περιφερειών ε, της Τσεχίας. σε ό,τι αφορά την οικονομική στήριξη και τον αριθμό των προγραμμάτων. Βλέπετε εδώ στο χάρτη ουσιαστικά την βελτίωση που έχει σημειωθεί και την αύξηση του αριθμού προγραμμάτων και την κατανομή τους ε, στις, τα έτη 2008, 2012 και 2016. Το 2016, για παράδειγμα, βλέπετε, είχαμε πάνω από 72.000 προγράμματα. Εδώ βλέπετε παραδείγματα αποτελεσμάτων, μια σύνοψή τους δηλαδή σε συγκεκριμένους ε, τομείς. Πάνω από 54.000 θέσεις εργασίας ε, δημιουργήθηκαν. Είχαμε σημαντικό αριθμό έργων ε, στο συνδρομικό δίκτυο, το οποίο είναι σημαντικό στοιχείο και για άλλες χώρες, γιατί η Τσεχία βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης και είναι και σημαντική χώρα και μετακόμισης και σε επίπεδο μικροπιστών επιχειρήσεων, παιδείας. Μπορείτε να τα δείτε αυτά τα στοιχεία και μετά. Σας φέραμε και ένα φυλάδιο και ένα βιβλίο μπορείτε να βρείτε δίπλα στην είσοδο. Και μπορείτε να τα διαβάσετε. Θα ήθελα να αναδείξω μια άλλη σημαντική διάσταση, οι δευτερεύουσες συνέπειες της πολιτικής συνοχής, από κλάδο σε κλάδο, αλλά όπως βλέπετε και στη διαφάνεια υπάρχουν τέτοιες ε, συνέπειες και για τις, από τις χώρες Βίζεγκρατ στις, ευρωπαϊκές, στις χώρες EU15. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τον αντίκτυπο της ε, πολιτικής συνοχής ε, σε όλες τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράδειγμα, βλέπετε ότι το ΕΕΠ των 12 χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια με βάση την πολιτική της συνοχής, ενώ στις χώρες Βίζεγκρατ είχαμε περίπου 77 δις ευρώ για τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 80% των κατανομών που επενδύουν οι 15 χώρες ε, στο κοινό προπολογισμό. Σε κάποιες χώρες είναι ακόμα παραπάνω. Από την μελέτη προκύπτει ότι έχουμε σημαντικά εξωτερικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την διαχείριση υδάτων, τις μεταφορές και την, τον περιορισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, εξοικονόμηση ενέργειας κτλ. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές δευτερεύουσες συνέπειες θετικές ε, της πολιτικής συνοχής, όχι μόνο για τις, ομάδες, τις χώρες της ομάδας Βίζεγκρατ, αλλά και για τα παλαιότερα κρατημέλη. Σε εξπόστα αξιολογήσεις μπορείτε να βρείτε και άλλα στοιχεία μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς έχει κατάσταση σήμερα στην Τσεχία. Εδώ έχει σημασία να δούμε μερικά στοιχεία λοιπόν και συνεχίζω με αυτά που είπε ο συνάδελφος ε, ε, γενικότερα. Για την Τσεχία λοιπόν πιο συγκεκριμένα. Σχεδόν όλες ε, οι προσφορές λοιπόν έγιναν δεκτές, πάνω από 530. 68,2% των ε, αιτήσεων που υπευλήθησαν και σχεδόν 80.000 ε, προγράμματα έχουν τώρα εγκριθεί. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, επιταχύνεται. Τους τελευταίους μήνες έχουμε λοιπόν μια επιτάχυνση κατά 10% σε όλα τα στάδια από την πρόσκληση υποβολή ενδιαφέροντο μέχρι το τελικό πρόγραμμα. Επομένω, ε, βρισκόμαστε σε σωστή τροχιά. Δύο λόγια τώρα για τις προγραμματικές ε, περιόδους. Καλό θα είναι να το αναφέρουμε εδώ, γιατί αν ε, στηρίξουμε αν συγκρίνουμε τι ε, δύο προγραμματικέ περιόδου, την προηγούμενη και την ε, τρέχουσα, τα πράγματα είναι διαφορετικά γιατί έχουμε διαφορετικέ πολιτικέ. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Ε, και έχουμε πολλά καινούργια στοιχεία, πολλέ νέε διατάξει και κανονισμού. Η τρέχουσα περίοδο έφερε μεταρρύθμιση και απαιτείται λοιπόν χρόνο για να προσαρμοστούμε. Πρέπει να μιλήσουμε εδώ για την αναγκαιότητα υιοθέτηση νέων στοιχείων όπω είναι ε, η εξάντε αιρεσιμότητα, το οποίο έχουμε υιοθετήσει μέχρι τα τέλη του 2016 και το πετύχαμε, το καταφέραμε αυτό. Στη συνοχή υπάρχει και ένα νέο στοιχείο της θεματικής συγκέντρωσης που τώρα μας δημιουργεί ορισμένες δυσκολίες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή γιατί υπάρχουν ε, δεκάδες ε, κανόνες σε ό,τι αφορά την κατανομή μεταξύ επιμέρους θεματικών στόχων υπάρχουν και νέες στοιχεία ό,τι φορά δημοσιονομικά μέσα και την ε, ε, διαδικασία ε, ορισμού. Και εδώ όμως τα καταφέραμε καλά ως Τσεχία και έχουμε και τις συστημικές αλλαγές όπως είναι το πλαίσιο επιδόσεων. Μπορεί να θεωρηθεί λοιπόν όλο αυτό σε ένα απαραίτητο βήμα προς τα μπρος Ταυτόχρονα όμως έχουμε και σημαντικά επίπεδα πολυπλοκότητας σε επίπεδο κανόνων και αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί στο μέλλον. Τώρα, ένα κρίσιμο παράδειγμα το οποίο δείχνει πόσο μας έχει επηρεάσει η, συνοχή, η πολιτική συνοχής. Το εύρος ε, της νομοθεσίας και των κατευθύνων γραμμών έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το 2013 Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πολύ σύνθετη η νομοθεσία και πλέον είναι αδύνατο να είναι κανείς ε, τέλειος και να τα αποκρίνεται γρήγορα. Συν ε, το σημείο εκκίνησης ε, καθυστέρησε αυτή την περίοδο εξαιτίας της καθυστερημένη υποβολή του, της τη νομοθετική νομοθετικής και μιας μακροχρόνιας διαπραγματευτικής περίοδου και αυτά λοιπόν πρέπει να επιληθούν πριν περάσουμε στην επόμενη περίοδο. Όμως ε, μάθαμε πράγματα από αυτή τη διαδικασία με τις νέες διατάξεις και έχουμε ε, επιφέρει κάποιες βελτιώσεις. Έχουμε ένα νέο ενοποιημένο ε, σύστημα μεθοδολογίας και παρακολούθησης, έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνου, έχουμε νέα μέτρα κατά της διαφθοράς. Αυτά σε στρατηγικό επίπεδο. Τώρα σε επιχειρησιακό έχουμε θέσει στόχους που συνδέονται με, τον, ε, με το ποσοστό των ε, προγραμμάτων που θα υιοθετούνται, περίπου 45% για φέτος. Πέρσι ο στόχος ήταν για τις ε, προσκλήσεις υποβολής ενδιαφέροντος στο 75%. Προσπαθούμε λοιπόν να συμπεριλάβουμε και αυτό το μέτρο. Ε, θέτουμε για κάποιες προβλέψεις πλέον και προσπαθούμε να καταλάβουμε αν θα υπάρχουν προβληματικά σημεία ή όχι. Αυτά είναι λοιπόν τα μέτρα που έχουμε υιοθετήσει αυτή την περίοδο και θα ήθελα να σταθώ και στην διασύνδεση μεταξύ των διευθυντικών ταμείων και άλλων μέσων Ε, έχουμε κάνει μια προσπάθεια λοιπόν να αναπτύξουμε συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων ΕΣΥΦ και άλλων ενωσιακών προγραμμάτων, αλλά δεν είναι εύκολο. Ε, υπάρχουν ε, θεσμικά, οικονομικά προσκόμματα, κάποιες φορές πρέπει για διαφορετικούς κόσμους. Προσπαθούμε λοιπόν να στηρίξουμε αυτές τις συνέργειες, γι' αυτό δημιουργήσαμε έναν μηχανισμό συντονισμού μεταξύ επιμέρους μέσων και Έχουμε ένα ευρύ φάσμα ε, φορέων όταν εξετάζουμε τις ε, αιτήσει, όχι μόνο με τα ταμεία ΕΣΥ, αλλά και με άλλα προγράμματα. Οι μηχανισμοί κεντρικής διαχείρισης θα πρέπει να τη διαχείριση από διαφορετικού φορεί. Ε, Επομένω, ε, πρέπει κάπω να διαβουλευτούμε και μαζί του για να δούμε τι μπορεί να γίνει καλύτερα. Εδώ βλέπετε ορισμένα παραδείγματα συνεργειών που διαμορφώνουμε ή βελτιώνουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ε, έρευνα, ανάπτυξη, εκπαίδευση για τον ορίζοντα 2020. και τώρα είμαστε κοντά στην υπογραφή της συμφωνίας και την υλοποίηση. Άλλο παράδειγμα είναι το ψηφιακό πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα, και καινοτομία για την ανταγωνιστικότητα και ε, το Clean Sky 2 Θέλουμε να βρούμε συνέργεια για το Clean Sky 2 λοιπόν μπορεί να ξεκινήσουμε διαφορετική διαδικασία για αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε λοιπόν παραδείγματα των όσων λαμβάνουν χώρα στην Τσεχία. Πληροφορίες έχουμε και σε ό,τι αφορά τους ε, περιορισμούς, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και πρέπει να πω ότι έχουμε αυτούς τους διαφορετικούς κόσμους για να υπάρξει προσέγγιση μεταξύ τους Πρέπει να εξετάσουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Χρειάζεται μεγαλύτερο συντονισμό, ίσως ε, και κατά τη απλούστευση ενδεχομένως. Υπάρχουν ε, διάφορα προσκόμματα και δυσκολίες, όπως είναι η εφαρμογή ορισμένων ε, κανόνων, κρατικέ ενισχύσει, επιλέξιμο κόστος, διαφορετικά συστήματα πληροφοριακά, και υπάρχει και μια έλλειψη επικοινωνία και πληροφόρησης μεταξύ των προγραμμάτων. Όλα αυτά πρέπει να λυθούν λοιπόν. Εάν θέλουμε να υπάρξει πραγματική διαμόρφωση συνεργειών μεταξύ των δύο μέσων. Είναι όμω διαφορετική και η φύση αυτών των ε, προγραμμάτων. Θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά και να μην υποστηρίζουν τα ίδια προγράμματα λοιπόν. Και εδώ αυτά τα μία είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης της περιφέρειας. Είναι μακροχρόνιος ε, στόχος, μακροπρόθεσμος δεν πρέπει να αλλάξουν οι στόχοι ε, σε σχέση με τώρα, θεωρούμε. Πρέπει να υπάρχει σαφής ε, αξιολόγηση των προτάσεων. Δεν έχουμε σωστή αξιολόγηση λοιπόν αυτών των ε, προγραμμάτων. Η προστατικότητα του Ταμείου, το, είναι σημαντική, καθώς και η κατανομή, η γεωγραφική κατανομή που ε, καταδεικνύει τεράστιες διαφορές αυτή τη στιγμή, γιατί οι παλαιότερες χώρες έλαβαν το 91% της οικονομικής στήριξης. Εντάξει, θα επιταχύνω. Τι θα γίνει στο μέλλον, λοιπόν. Εμείς ε, μάθαμε ότι είχαμε να μάθουμε, έχουμε αποκτήσει τις απαραίτητε γνώσεις, ξέρουμε ποιες είναι οι προκλήσεις, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και δηλώνουμε και την δέσμευσή μας να αλλάξουμε το σύστημα, το οποίο μπορεί να σημάνει και την απλούστευση στο μέλλον. Να σταθώ σε τρία-τέσσερα στοιχεία, τα οποία είναι σημαντικά για το μέλλον και για την Τσεχία αλλά και ευρύτερα. Χρειαζόμαστε ένα στρατηγικό όραμα για το 2030, συγκεκριμένου στόχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μα. Να δούμε πού οδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τώρα μεταρρύθμιση τη πολιτική συνοχή. Παρά ότι δεν έχουμε ξεκαθαρά στοιχεία για κάποια από τα νέα δεδομένα τη μεταρρύθμιση, βλέπουμε όμω μια συνέχεια, να μην έχουμε μια ριζική τομή σε στρατηγικό επίπεδο. Αυτό είναι σημαντικό προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι η τρίτη περίοδος για μας. Κάποιες φορές νιώθουμε ότι βρισκόμαστε πάντα ξεκινάμε από το μηδέν με νέε διατάξει, νέου κανόνε. Η ε, ε, επιμερισμένη διαχείριση είναι βασική αρχή τη πολιτική συνοχή. Θα πρέπει λοιπόν να την ε, συνεχίσουμε να την υιοθετούμε, να την εφαρμόζουμε αλλά να την βελτιώσουμε. Σημαντική είναι και η απλούστευση. Πρέπει να έχουμε νέο πλαίσιο βάση τη εμπειρία με γνώμονα του στόχου αλλά να μην παραλύσουμε την πολιτική συνοχή από έναν υπερβολικό αριθμό ε, κανόνων και περιορισμών. Νομίζω ότι υπερεύει το χρονικό μου όριο. Δύο πράγματα θέλω μόνο να αναφέρω. Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι εκ των προτέρων και το, η νέα δέσμη για το νέο ΠΔΠ θα πρέπει ε, να είναι έτοιμη το στόμα δυνατόν. Το αργότερο μέχρι το Μάιο του 2018, ιδάλλως ε, θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα που είχαμε και στο παρελθόν. Και στην τελευταία διαφάνεια βλέπετε πώς μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από την Τσεχία σε ό,τι φορά τα αριθμητικά στοιχεία. Και έχετε στην είσοδο και ορισμένα φυλάδια, όπως σας είπα και προηγουμένως. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σκόνα, για την παρουσίασή σας, ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη και διεξοδική, για την Τσεχία. Να δώσουμε τώρα το λόγο. Κύριε Μάνκα, θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με τις δύο αυτές παρουσιάσεις ε, που ακούσαμε. Ε, στην πρώτη ε, έγινε λόγος για, την, για τον συνδυασμό των ΕΔΕΤ με το ΕΦΣΙ μεταξύ άλλων και αναφέρθηκε επίσης και το γεγονός ότι η Σχετική Επιτροπή ήταν κάθετα αντίθετη σε αυτή την ιδέα. Στην δεύτερη τώρα παρουσίαση ακούσαμε ε, πως ε, ε, ενδεχομένως δεν είναι πάντοτε θεμητό το να μετακινούνται ή να μεταφέρονται κονδύλια από τον ένα μηχανισμό στον άλλον. Με βάση τώρα την πρόταση όμπνιμπους της Επιτροπής, εκείνο που προβλέπεται είναι ότι τα κονδύλια, τα εκάστοτε κονδύλια θα μπορούν να κατευθύνονται προς το κράτος μέλος εκείνο το οποίο τα χρειάζεται. Δηλαδή, εάν περισσεύουν τρόπο την, ε, ε, κονδύλια σε ένα κράτος μέλος από ένα ταμείο, τότε μπορούν να ανακατευθυνθούν τα εν λόγω κονδύλια σε άλλους τομείς αλλά της ίδιας ε, περιοχής. Ενδεχομένως η λύση λοιπόν η οποία προτείνεται με, το, με την πρόταση Omnibus να έχει κάποιο νόημα. έχει δημιουργηθεί, δηλαδή έχει προταθεί αν θέλετε αυτή η, η, λογική του να επιστρέφουν ουσιαστικά τα κονδύλια εκεί που πρέπει και μπορούμε ενδεχομένω ε, για να το επιτύχουμε να ε, αξιοποιήσουμε τους κανόνες που ήδη ισχύουν στο πλαίσιο του Ταμείου Στρατηγικών ε, Επενδύσεων. Ίσως λοιπόν η μεταφορά των λόγω κανόνων και στα υπόλοιπα ε, ταμεία θα είχε νόημα. Ακριβώς στο πλαίσιο και της πρότασης Όμνιμπους. Τώρα, σε σχέση με τα υπόλοιπα ζητήματα που αναφέρθηκαν στις δύο παρουσιάσεις. για παράδειγμα η απλούστευση των κανόνων ε, όταν έχουν εξοικειωθεί πολύ καλά τα κράτη-μέλη με τους εν λόγω κανόνες. Ε, προφανώς κανείς δεν θέλει να περιπλέκουμε περαιτέρω τα πράγματα, αλλά αν δούμε το τι συμβαίνει στην πράξη, όλες ε, οι κυβερνήσεις ε, ειδικότερα δηλαδή των δικαιούχων κατομελών που απορροφούν τα περισσότερα κονδύλια, αναφέρουν ακριβώς ε, το, το πρόβλημα που δημιουργεί το διοικητικό άχθος, ε, αναφέρουν επανειλημμένα την ανάγκη δηλαδή για περαιτέρω απλούστευση, η οποία με τη σειρά της μπορεί να επιτρέψει εξοικονόμηση κονδυλίων, για παράδειγμα μέσω διεξαγωγής λιγότερων ελέγχων, επιθεωρήσεων και ούτω καθεξής. Δηλαδή πρόκειται για λογικά στοιχεία ε, τα οποία όλοι μας μπορούμε να τα σκεφτούμε. Δηλαδή δεν μπορούν ε, ε, όλοι οι δήμοι και οι κοινότητες να ε, συνεχίσουν να υποβάλλονται σε πλήρης ε, ε, ελέγχους ανά δύο ή τρία έτη. Επίσης έγινε μια αναφορά στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο επίπεδο για παράδειγμα της εκτέλεσης των, γενικών, των έργων αυτών των ταμείων, ότι δηλαδή είναι αργοί οι ρυθμοί, σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν και επαρκή έργα τα οποία συμμετέχουν, σε άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό για τη διαχείριση των λόγω έργων αλλά θα, ήθελα να σας υπενθυμίσω πως ε, ε, έγινε μια, εκπονήθηκε μια μελέτη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις της πληρωμές και ίσως λοιπόν η δημοτόπιση αυτού του είδους των καθυστερήσεων να μπορούσε να βοηθήσει. Εγώ δηλαδή όταν ήμουν δήμαρχος στη δική μου πόλη πραγματικά είχα διαπιστώσει το πόσο αρνητικό ε, είναι ε, αυτό το σύστημα. Δηλαδή, οι συνάδελφοί μου μου λέγανε ότι δεν θα ε, βασιζόμαστε σε συγχρηματοδότηση, για παράδειγμα, για την οικοδόμηση γεφυρών, γιατί ακριβώ καθυστερεί η εκταμείευση των σχετικών κονδυλίων έως και δύο χρόνια. Ίσως λοιπόν αυτό το ζήτημα τη αρκοπορία στι πληρωμέ μπορεί να βοηθήσει στην εξήγηση του γιατί υπάρχει γενικότερα καθυστέρηση στην εκτέλεση του προπολογισμού. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Όλμπερτ έχει στήσει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ακούσουμε μάλλον και τους επόμενους ομιλητές, φαντάζομαι. Αλλά να πω μια γνώμη για τα όσα ακούσαμε μέχρι τώρα. Η συζήτηση που λαμβάνει τώρα στην Επιτροπή Ρέντζη, λοιπόν, πώς έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή. Έχουμε βέβαια το πρώτο ερώτημα που θέσαμε και στον εισηγητή. Το ΕΦΣΙ, ποιο σκοπό εξυπηρετεί τελικά. Ποιο είναι ο στόχο, το θυμάμαι τότε ότι υποτίθεται ότι αφορούσε τα πλέον επικίνδυνα και ρηψοκίνδυνα προγράμματα. Εάν κάτι είναι πολύ επικίνδυνο για το ΕΦΣΙ, τότε ποιο είναι ο σκοπό του ΕΦΣΙ. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα για μένα κατανοώ ε, το κριτήριο του τριπλού α για τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες Επενδύσεων, αλλά μου είπαν ότι το, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων απορρίπτει το ΕΦΣΙ γιατί είναι πολύ ρίψο Αλλά ποιο είναι ο σκοπό του ΕΦΣΙ τελικά. Σήμερα όμω συζητούμε την σύνδεση μεταξύ ε, του ΕΦΣΙ και των υπολείπων ε, ταμείων κτλ. Επομένω, θέλουμε εμεί να ενισχύσουμε τη συμπληρωματικότητα ή να βρούμε μια στρατηγική ε, διεξόδου για τα κονδύλια που δεν έχουν δαπανηθεί να τα στρέψουμε στο ΕΦΣΥ. Γι' αυτό είναι το πρόβλημα με το Omnibus, γιατί εκεί η ιδέα της συμπληρωματικότητα που υπάρχει είναι σωστή, όμως ε, προτείνεται χρήματα της συνοχής να περάσουν στο ΕΦΣΥ. Και αυτό είναι πραγματικά αυτή η ε, στρατηγική διεξόδου. Όσα δεν δαπανώνται να τα δίνουμε στο ΕΦΣΥ. Το ακόμα πιο σημαντικό, ποιο είναι το πρόβλημα μεταξύ του ΕΣΥΦ και του ΕΦΣΥ. Είναι διαφορετικές οι προϋποθέσεις, διαφορετικά τα κριτήρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν μπορεί να εξετάσει συγκρίσιμες ε, προδιαγραφές, για παράδειγμα κρατικές ενισχύσεις, γιατί εμείς θα δούμε το φαινόμενο να φεύγουν κάποιοι από την πολιτική συνοχή και να πηγαίνουν στο ΕΦΣΙ, γιατί θα είναι πιο εύκολο. Όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, θα είναι πιο εύκολο δηλαδή γραφειοκρατικά και διαδικαστικά. Αυτό αναφέρει και ο εισηγητή. Είναι το πρόβλημα που είχαμε και στην Επιτροπή Ρέτζη σήμερα. Το θέμα του Συμφώνου Σταθερότητα έναντι πολιτική συνοχή. Έχουμε του ίδιου κανόνε για τα ΕΣΥΦ και το ΕΦΣΙ. Στο ένα έχουμε επιμερισμένη διαχείριση, στο άλλο όχι. Αν έχουμε λοιπόν μεικτή διαχείριση, άμεση διαχείριση ή διαχείριση ΕΤΕΠ που είναι ιδιαίτερη, μπορούμε να διαβιβάσουμε κονδύλια από το ένα στο άλλο που έχουν τελείως διαφορετική μεθοδολογία. Αυτό πρέπει να απαντηθεί λοιπόν. Ίσως το κάνουν οι δύο επόμενοι ομιλητέ. Υπάρχει μία σαφής εργαλειοθήκη. Αν κάποιος θέλει να ελοποιήσει ένα πρόγραμμα, πού είναι τα χρήματα. Τα χρήματα τα έχει είτε το ΕΦΣΙ είτε τα ΕΣΥΦ. Υπάρχουν κανόνες. Είναι σαφείς ή μπορεί κανείς να πάει πρώτα στο ένα ή στο άλλο. Διαφορετική συνοχή ε, στο ένα ή στο άλλο μέσο, οπότε επιλέγει. Εγώ διαφωνώ. Δεν νομίζω ότι είναι μια σωστή προσέγγιση. Πρέπει να έχουμε μια ξεκαθαρή εικόνα. Ίσως δεν είμαι σωστά ενημέρωμένο αλλά πιστεύω πραγματικά ότι χρειάζεται μια ξεκάθαρη απάντηση, γιατί δημιουργήσαμε αυτά τα μέσα και πρέπει ε, να είναι σαφές για τους δικαιούχου πώς θα πρέπει να τα αξιοποιήσουν και όχι μόνο να σκέφτονται το τριπλό α. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Όλπριχτ. Δεν ξέρω τώρα τι πρέπει να κάνω. Ίσως το καλύτερο θα ήταν να επιτρέψουμε Θέλετε να θέσετε μια ερώτηση τώρα, θα κάνουμε τη συζήτηση τώρα, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει χρόνος μετά να δώσουμε το λόγο στους άλλους δύο μιλικέτες. Προτείνω επισήμως να περιμένουμε τις δύο τελευταίες παρουσιάσεις, μπορεί να απαντήσουν στις ερωτήσεις που ετέθησαν. Ε, να δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στον κύριο Νούνιες Φερέρ, ο οποίος είναι ανεξάρτητος ε, σύμβουλος του Κέντρου ε, Ευρωπαϊκών πολιτικών μελετών. Ναι, εργάζομαι ε, για το ε, κέντρο αυτό και είμαι και σύμβουλος ε, που σημαίνει βέβαια ότι μου αρέσει να ασχολούμαι και με πραγματικά έργα, δηλαδή να βλέπω πώς είναι η πραγματική τους ελοπίση. Αυτό δηλαδή μου δίνει και μια εμπειρία στο πώς λειτουργούν στην πράξη τελικά τα ταμεία. Άρα λοιπόν αυτό που μου ζητήθηκε είναι να δώσω κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν. Θα αναφερθώ και στα όσα υπόθηκαν, αλλά εντάξει, μία απάντηση ε, εντός 10 λεπτών δεν είναι ποτέ δυνατόν να δοθεί. Έχω προετοιμάσει λοιπόν μία δεκαλεπτή παρουσίαση και έχουμε δημοσιεύσει από την πλευρά του ΣΕΠΣ μία δημοσίευση FC2-0, ε, δηλαδή η δεύτερη εκδοχή. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που μπορώ να πω στον κύριο Όλμπριχτ είναι ότι δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιε επιμέρου απαντήσει, αλλά δεν υπάρχει μια πλήρη ε, γενική απάντηση. Ε, λοιπόν, ε, ω προ το τι χρειαζόμαστε, εγώ διάβασα την πρόταση. Ο είναι κάπω ε, υπερβολικά περεκτική, αν θέλετε λίγο. Είναι υπερβολικά όμνικα, τη δική μου άποψη. Ε, εντάξει, εμεί οι ερευνητέ ούτω ή άλλω δεν μα αρέσει πολύ να διαβάζουμε νομοθεσία. Ε, ποια είναι σε κάθε ε, περίπτωση τα θεμελιώδη ζητήματα. Σε αυτό θέλω να εστιάσω. Γιατί υπάρχουν δηλαδή τα ΕΔΕΤ, γιατί υπάρχει το Ταμείο για τις ε, Στρατηγικές Επενδύσεις και πώς θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Γιατί αν διαβάσουμε όλη την νομοθεσία, πραγματικά θα ε, διαπιστώσουμε ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Ε, γιατί ε, αν συγκρίνουμε δηλαδή το τι προτείνεται τώρα σε σχέση με την ενδιάμεση αναθεώρηση και τις χειρές προτάσεις του 2010, θα δούμε ότι πραγματικά εδώ πραγματικά υπάρχει πρόοδος. Παρ' όλα αυτά αφήνουμε μία σειρά από κενά και υπάρχουν απλουστεύσεις οι οποίες τελικά θα οδηγήσουν σε περισσότερα προβλήματα. Και θα εξηγήσω σε λίγο το τι εννοώ. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα προπολογισμό ο οποίο θα ανταποκρίνεται στι σημερινέ ανάγκε. Ε, αυτό είναι βασική ανάγκη. Χρειαζόμαστε μια ε, ολοκληρωμένη ένα ολοκληρωμένο προγραμματισμό και αυτό γίνεται όλο ένα και πιο σημαντικό. Δηλαδή θα πρέπει, αφού έχουμε όλο ένα και περισσότερα ταμεία και περισσότερα εργαλεία, να, να συντονίζουμε καλύτερα μεταξύ μα εργαλεία σε ό,τι αφορά δηλαδή την καταπολέμηση τη ανεργία, την ε, αύξηση τη επιχειρηματικότητα και ό,τι καθεξή. Αυτή η περιεκτική, αν θέλετε, ολοκληρωμένο ο προγραμματισμό δημιουργεί προβλήματα για διάφορε διοικητικέ αρχέ οι οποίε είχαν συνηθίσει στην εξειδίκευση και που πρέπει τώρα να περάσουν σε πιο ολοκληρωμένε ακριβώ αντιμετωπίσει. Αυτό ισχύει για όλου του τομεί, όχι μόνο για το τομέα τη δημόσια χρηματοδότηση. Χρειαζόμαστε επίση καινοτόμε λύσει, γιατί βρισκόμαστε σε έναν ε, ταχύω μεταβαλλόμενο ε, καινοτόμο κόσμο. Οπότε θα πρέπει να αναπτύξουμε τις κατάλληλες λύσεις παρά την υφιστάμενη γραφειοκρατία. Τι σημαίνει αυτό. Χρειαζόμαστε καινοτόμε ε, δημόσιες συμβάσεις, χρειαζόμαστε συνδυασμό των ενισχύσεων των χρηματοδοτικών εργαλείων και του ιδιωτικού τομέα. χρειαζόμαστε και αυτό είναι απαραίτητο παντού, δηλαδή είναι κάτι που συμβαίνει ένα κίνημα, αν θέλετε, ένα φαινόμενο που ε, παρατηρείται παντού αυτή η καλύτερη, δηλαδή ο καλύτερο συνδυασμό των χρηματοδοτικών εργαλείων του ιδιωτικού ε, τομέα. Ταυτόχρονα χρειαζόμαστε περισσότερη κοινωνική καινοτομία, δηλαδή ε, εάν γίνεται μια πρωτοβουλία χωρί όμω να υπάρχει συμμετοχή των πολιτών, ουσιαστικά οδηγούμαστε σε απώλειε γιατί ο κόσμο ουσιαστικά δεν υιοθετεί, αν θέλετε, τη νέα λύση. Ε, αυτό, για παράδειγμα, αφορά σε μεγάλο βαθμό την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα, αφορά επίση το τομέα των μεταφορών. Χρειαζόμαστε δηλαδή καινοτομίε οι οποίες ε, να, είναι, να οδηγούν σε, σε κοινωνική μεταβολή και ταυτόχρονα χρειαζόμαστε και πρωτοβουλίες οι οποίες επιτυχάνουν ταυτόχρονα διαφορετικούς, πολλούς διαφορετικούς στόχους. Ε, και είναι δύσκολο να επιτυχάνουμε διαφορετικούς στόχους και να επιτυχάνουμε και κοινωνική ε, καινοτομία. Και επίσης χρειαζόμαστε να ξεφύγουμε λίγο από τις ε, γκρίζες επενδύσεις τις οποίες παραδοσιακά επενδύει ο δημόσιο τομέα, και να γίνει ένας ε, στρατηγικός επενδυτής για παράδειγμα ε, το δημόσιο. Δηλαδή αντί να προβαίνει για παράδειγμα στην οικοδόμηση γεφυρών και να λέει ότι εντάξει τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει ο ιδιωτικό φορέα, το δημόσιο καλείται από εδώ και στο εξή να αποτελέσει έναν ε, κοινωνικό επιχειρηματία, αν θέλετε, social entrepreneur. Και ακριβώ εδώ εντοπίζονται και κάποια από τα σημαντικότερα προβλήματα. Ποια είναι λοιπόν τα θεμελιώδη προβλήματα σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το πιο σημαντικό πρόβλημα, ειδικότερα του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αν δεν υπάρχει ε, εμπιστοσύνη τότε ε, δεν παίζει ρόλο το πόσο μεγάλη απλούστευση θα κάνουμε γιατί πάλι θα περιπλέξουμε τα πράγματα. Γιατί ε, αν υπάρχουν ένα σώρο από φορεί και κράτη-μέλη τα οποία λένε τι κάνετε εδώ, θέλουμε μια εξαίρεση εδώ, θέλουμε μια εξαίρεση εκεί, τότε ουσιαστικά περιπλέκουμε τα πράγματα περισσότερο. Και δεν υπάρχει τίποτα ε, πιο περίπλοκο από έναν κανόνα με πολλέ εξαιρέσει. Και αυτό το γνωρίζουμε και από τη γαλλική γλώσσα, αν θέλετε. Εντάξει, αστείευομαι τώρα, αλλά πραγματικά, εάν η εξαίρεση γίνεται ο κανόνα σε αυτέ τι περιπτώσει, τότε έχουμε πραγματικά προβλήματα. Και αυτό ακριβώ συμβαίνει με τα χρηματοδοτικά του μάτια τη Ένωση. Από εκεί και μετά έχουμε υπερβολική περιπλοκότητα. Δηλαδή έχουμε ψηλό διοικητικό άκθο και μετά και ε, ε, ε, υπερβολική εστίαση στην, ε, στις διαδικασίες. Ε, δηλαδή είχε ε, εδώ και κάποια χρόνια υιοθετηθεί από την Επιτροπή η, στάση του ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δρά ως φορέας διαχείρισης των ταμείων. Αλλά αυτό οδήγησε τελικά στο ουσιαστικά σε εκ προτέρων προστασία των οικονομικών τη συμφερόντων, ακριβώ επειδή δεν υπάρχει ανάληψη των ευθυνών μετά την υλοποίηση των προγραμμάτων από τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, εάν δεν μπορεί να, ε, ε, να καταστήσει υπόλογα τα κράτη-μέλη, η Επιτροπή τι θα κάνει, ουσιαστικά προσπαθεί εκ των προτέτων να ε, διασφαλίσει τα συμφέροντά της. Δηλαδή, Ακριβώ επειδή δεν υπήρξε αυτή η απόδοση των ευθυνών στα κράτη-μέλη, οδηγηθήκαμε στο, στη σημερινή κατάσταση. και επίση, αν διαβάσουμε και διάφορε εκθέσει ό,τι αφορά για παράδειγμα τους πολλαπούς ελέγχους, ε, την, ε, της κατεξουσιοδότηση ε, νομοθετικές πράξεις, θα διαπιστώσουμε ότι πραγματικά δημιουργούμε περισσότερη περιπλοκότητα μέσω μιας υποτιθέμενης απλούστευσης. Τώρα, ε, ε, διαπιστώνουμε λοιπόν με βάση αυτού του στόχου ότι παρότι φαίνονται παράλογοι, υπάρχει μια λογική που έχει οδηγήσει στην ύπαρξή του. Από εκεί και μετά λοιπόν, μετά από αυτή την περιπλοκότητα, έχουμε και τον κατακαιρματισμό. Δηλαδή, έχουμε μια σειρά από διαδικασίε που ακολουθούν διάφορε γενικέ διευθύνσει για τα διαφορετικά προγράμματα. Ε, έχουμε μια σειρά από διαφορετικά έντυπα υποβολή αιτήσεων. Έχουμε διαφορετικέ υποβολέ εκθέσεων. Διαφορετικού ελέγχου για παράδειγμα, διάβαζα ε, σχετικά με ένα έργο στις ε, κάτω χώρε όπου οι αρμόδιοι του έργου έπρεπε να συνεργάζονται με τρεις γενικές ε, διευθύνσεις και να υποβάλλονται σε τρεις διαφορετικούς ελέγχους. Γιατί αυτό συμβαίνει συχνά. Δηλαδή, αναλαμβάνει κανείς ένα συνδυασμένο τέτοιο έργο διατομιακό, αλλά τελικά βρίσκεται υπόλογο σε τρει διαφορετικέ γενικέ διευθύνσει, Πρέπει να υποβάλει τρει εκθέσεις, να υποβάλλεται σε τρει έλέγχου. Έχουμε λοιπόν ταυτόχρονα το καταγερματισμό των ταμείων σε ό,τι αφορά τον ε, εκ των προτέρων καταμερισμό των ταμείων, την ε, επιλεξιμότητα και ούτω καθεξής. Τι σημαίνει αυτό, ότι συχνά δηλαδή οι διαδικασίε οι οποίες ισχύουν ήδη είναι παροχημένε σε σχέση με όσα θέλουμε να επιτύχουμε ε, σήμερα δηλαδή. Η επιλεξιμότητα των σχετικών μέσων δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Για παράδειγμα στον τομέα της γεωρίας, για παράδειγμα επειδή υπήρξε μια ιστορική απόδοση το 2009 ή το 2005, ε, βασιζόμαστε πάντα στο κατακεφαλήν ΑΕΠ, αλλά για παράδειγμα παραβλέπουμε μια ε, σειρά από περαιτέρω τομείς, για παράδειγμα όπως το εισόδημα, την ε, ε, οικονομική κατάσταση και ούτω καθεξής. Ε, σε, συχνά δηλαδή αυτό που έχει μείνει ιστορικά, απομείνει αν θέλετε ιστορικά στον προπολογισμό, ε, μας οδηγεί στο να μην ανταποκρίνεται ο προπολογισμό στις ανάγκες. Αφού σας παρουσιάσα λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα, σας εξηγώ το τι συμβαίνει γενικά, ότι έχουμε υψηλότερη περιπλοκότητα και αλληλεπικάλυψη ακριβώς μεταξύ των διαφορετικών ε, χρηματοδοτικών εργαλείων, των διαδικασιών, των ελέγχων και ούτω καθεξής. Έχουμε την κοινή χρηματοδότηση όπου βλέπετε εδώ ε, στη μέση, δηλαδή ε, υποδομές, υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και καινοτομία. Αλλά από εκεί και μετά έχουμε και τα κεντρικά ταμεία, δηλαδή την ε, διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη, το ΕΦΣΥ, μετά έχουμε τη ΣΥΝΟΦΗ για την υποστήριξη των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το COSME και αυτό για την υποστήριξη της κοινοτομία στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και ε, το ΕΦΣΥ για την υποστήριξη και αυτό της κοινοτομία στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αν λοιπόν ρίξει μια ματιά κανεί σε όλο αυτό το σύστημα, να ρωτιέται ποιο είναι αρμόδιο γιατί και τι κάνει. Και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε για την επόμενη αναθεώρηση. Ας δούμε λοιπόν, ε, μου μένει άλλο ένα λεπτό, ας δούμε λοιπόν τι ε, συμβαίνει στο επίπεδο της ενδιάμεσης ε, αναθεώρησης. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι λοιπόν σε ό,τι αφορά την, ε, το flat rate financing, αυτή τη χρηματοδότηση του ενιαίου ποσοστού. Ναι, ε, είναι θετική ω πρόταση, αλλά θα ισχύει ακριβώ στι περιπτώσει όπου υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη και θα προβλέπονται εξαιρέσει, ε, κατεξουσιοδότηση νομοθεσία και ούτω καθεξή. Τι σημαίνει αυτό, Αυτό θα σημαίνει υψηλότερα ποσοστά λάθου και θα αρχίσει ο τύπο να λέει ότι είστε διαφθαρμένοι και ούτω καθεξή. Δηλαδή υπάρχει μια καλή ιδέα που εφαρμόζεται και μετά προβλέπουν ταυτόχρονα κατεξουσιοδότηση πράξη που ε, επιτρέπουν ουσιαστικά στην Επιτροπή να πάρει κλίνη από αυτόν τον κανόνα, από αυτό το σύστημα. Ε, από εκεί και μετά. Ο προπολογισμό που θα βασίζεται στι επιδόσει είναι μια καλή ιδέα και νομίζω πω θα εφαρμοστεί, αλλά νομίζω πω αρχικά είχε προβλεφθεί ε, ως αντίβαρο αν θέλετε ή ω εναλλακτική λύση στην απλούστευση. Εδώ τι λέμε τώρα, θα ε, προβούμε σε περαιτέρω απλούστευση και μετά θα έχουμε και, την, ε, και το παλιό σύστημα σε ό,τι αφορά δηλαδή την την εστίαση στις επιδόσεις. Ουσιαστικά δηλαδή θα παραμείνει και το άχθος από το παλιό σύστημα και θα προσθέσουμε περαιτέρω άχθος. Και εδώ επανέρχομαι βέβαια στο, σύστημα, στο, συγγνώμη, στο ζήτημα της εμπιστοσύνης. Δηλαδή αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιο προπολογισμό που βασίζεται στι επιδόσεις. Μετά σε ό,τι αφορά την, την απλούστευση και το και την εναρμόνιση και πάλι εδώ αναφέρομαι στο ζήτημα της εμπιστοσύνης. Δεν ξέρω δηλαδή εάν θα υπάρξει τελικά, ένα ενιαίο σύστημα που θα εφαρμόσετε ως ε, τέτοιο. Σε ό,τι αφορά το συνδυασμό ΕΔΕΤ ε, και ΕΦΣΙ ναι, ε, ειδικότερα σε ορισμένε περιπτώσει σε Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη, σε συνδυασμό με το ΕΦΣΥ για παράδειγμα, μπορεί καλά να λειτουργήσει. Αλλά εκεί βέβαια τίθεται το ερώτημα του ποιο θα είναι εκείνο ο οποίο θα δίνει τι εγγυήσει, ποιο ταμείο. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, συμπληρωματικότητα και τι συνέργειε, υπάρχει ο μεγάλο κίνδυνο κατακαιρματισμού των σχετικών κανόνων και διαδικασιών μεταξύ γενικών διευθύνσεων και αυτό ο κίνδυνο παραμένει γιατί βέβαια οι, αυτοί οι φορεί, αν θέλετε, γενικέ διευθύνσει δεν αλλάζουν τόσο εύκολα. Μετά σε ό,τι αφορά την ευελιξία, φοβούμε ότι θα κάνουμε το ίδιο ε, πράγμα που γινόταν μέχρι τώρα. Δηλαδή κάποια στοιχεία που έχουν χαμηλή προστιθέμενη αξία να απορροφούν ουσιαστικά μέρος των κονδυλίων ε, από στοιχεία υψηλή προστιθέμενη αξία. Δηλαδή, ε, να παίρνει κανεί, για παράδειγμα, από το Horizon ή από το κόσμο κάποια κονδυλία και να κατευθύνει αλλού, που δεν έχουν τόσο μεγάλη χρησιμότητα. Τέλο, σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά προτινόμενα ε, επιστηματικά ταμεία, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο αποδυναμώνουμε την ενότητα του προπολογισμού και μειώνουμε και την ε, το επίπεδο της χρηστής διακυβέρνησης. Ε, ε, συνολικά λοιπόν θεωρώ πως πραγματικά θα υπάρξει ένας καλύτερος ε, προπολογισμό με βάση τις νέες προτάσεις αλλά υπάρχουν ακόμα πολύ σημαντική κίνηση. Θα πρέπει να κινηθούμε προς έναν ε, απλουστευμένο προπολογισμό και η έμφαση δεν πρέπει να δοθεί τόσο στα διαφθορτικά και επενδυτικά ταμεία. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος, ένα ενιαίο κονδύλια, θέλετε, ένα ενιαίο κομπανάς ο οποίος θα επιτρέπει ακριβώς τη μεγάλη, ε, τον μεγάλο καταμερισμό των σχετικών κινδύνων, των χρηματοδοτικών κινδύνων. Δηλαδή, η εγγύηση ούτω ή, άλλω θα πρέπει να υπάρχει, είτε αυτή προέρχεται από το Ταμείο συνοχή ή οποιοδήποτε άλλο ταμείο, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν το κονδύλι είναι κοινό, έχουμε ακόμα καλύτερη, ακόμα υψηλότερη κατανομή των σχετικών κινδύνων. Για παράδειγμα, εάν έχουμε διάφορε περιοχέ οι οποίες ε, συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα, αν προσθέσουμε και για παράδειγμα περιοχέ τη Γερμανία κατευθείαν μειώνουμε τον γενικότερο ε, κίνδυνο τη υλοποίηση αυτού του έργου. άρα λοιπόν έχουμε στο πλαίσιο τη ενδιάμεση αναθεώρηση κάποιε βελτιώσει, αλλά δεν είναι ιδανικά τα πράγματα. Θέλουμε δηλαδή να έχουμε πιο απρόσκοπη χρήση των επιχορηγήσεων, θέλουμε καλύτερο καταμερισμό, δηλαδή ο οποίο θα βασίζεται στι ε, εκαστοτε ανάγκε. Χρειαζόμαστε να μειώσουμε την ε, αυξανόμενη περικλουπλοκότητα των ε, σχετικών χρηματοδοτικών εργαλείων, γιατί βέβαια θα πρέπει να εστιάζουμε και στη ζήτηση, όχι μόνο στου στόχου του προπολογισμού. Και από εκεί και μετά επανέρχομαι στο ζήτημα τη γενικότερη απλούστευση, δηλαδή σημεία ενία εξυπηρέτηση ε, μία ενιαία διαδικασία υποβολή αίτηση, ένα ενιαίο έλεγχο. Δηλαδή, όταν κάποιο είναι δικαιούχο, ε, θα πρέπει όχι να τον απασχολεί το πώ θα λάβει τη χρηματοδότηση από τα διαφορετικά ταμεία. Εκείνο που θα πρέπει να τον ενδιαφέρει είναι το να προτείνει ένα ποιοτικό ε, έργο. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νιούνιες Φερέρ για αυτή την παρουσίαση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ζουλιάν Γουατρί από την ε, εταιρεία επενδύσεων της Τρίτης Βιομηχανικής Επανάστασης. Να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ που δώσατε και λίγο χρόνο και σε εμά. Θα σας μιλήσω πολύ σύντομα, αν θέλετε να βάλετε και τις διαφάνειες, ε, για την ε, περιοχή της Γαλλίας η οποία θέλει να ξεκινήσει την τρίτη βιομηχανική επανάσταση. Έχασε τη δεύτερη και εδώ και κάποια χρόνια, εδώ και τρία χρόνια πιο συγκεκριμένα, αποφάσισε να αναλάβει τα ενία και να ε, επικεντρωθεί στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε την τρίτη βιομηχανική επανάσταση, την έννοια. Ένας οικονομολόγος, ο Τζερέμι Ρεύκιν, ε, αναφέρθηκε σε μια οικονομία η οποία θα μπορούσε να αναπτυχθεί σήμερα χάρη σε μια ε, οικονομία χωρίς χρυσή άνθρακα και επομένως πιο φθηνή. Στην συγκεκριμένη περιοχή, που είναι μια περιοχή χωρίς άνθρακα, Carbon Zero Region, μία από τις πρωτοβουλίες λοιπόν της Region France ήταν πριν από 1,5 χρόνιο να ξεκινήσει το Ταμείο για την τρίτη βιομηχανική επανάσταση. Πρόκειται για το CAP3RI. Πρόκειται για ένα ταμείο το οποίο υποστηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, χάρη λοιπόν στο Ταμείο Ευρωπαϊκής, Ένωσης, ε, Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης, το ΦΕΝΤΕΡ και το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το Ταμείο Juncker. Πρόκειται για ένα ταμείο το οποίο βασίζεται ε, στην ενεργειακή ε, πτυχή και θέλει να έχει μια οικονομία χωρίς άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τα πάντα διαπιστώνονται από το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιες ελλείψεις για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και επομένως θα πρέπει να υπάρχει σύσταση ενός ταμείου, ενός ταμείου το οποίο θα πρέπει να χρηματοδοτήσει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις καινοτόμες επιχειρήσεις, ε, νεοφυείς επιχειρήσεις λοιπόν οι οποίες ε, δοκιμάζονται και αποδεικνύουν την αξία του συνεχώς και επομένως προσπαθούμε να έχουμε χρηματοδότηση και αυτών. Και χάρη στη μελέτη αυτή διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται και τεχνική υποστήριξη η οποία θα επιτρέψει να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέα προγράμματα. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Όσον αφορά το θέμα του διαχειριστή του Ταμείου. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015, πριν 1,5 χρόνο λοιπόν, και μία από τις ε, προτεραιότητες ήταν ότι ο διαχειριστής θα πρέπει να επενδύσει 5 εκατομμύρια ευρώ ε, για το χρηματοδοτικό αυτό μέσο ο επιτυχής υποψήφιος ήταν η North Capital Partners ε, σε συνεργασία με την Φινόπρα και η, επίσης επένδυσε και η Crédit Αγκρικόλ ε, της Βόρειας Γαλλίας. Και γιατί αυτό, γιατί ήταν ε, ο με το μετοχός, επομένως είχε ένα ποσοστό και τα υπόλοιπα αντιστοιχούν σε ένα ταμείο επενδύσεων που λέγεται... Capital και αυτοί διαθέτουν αρκετές επενδύσεις στην περιοχή της Γαλλίας. Και έχουμε και ένα ταμείο επενδύσεων το οποίο χρηματοδοτείται και από δημόσια κονδύλια ε, μέσω του ΕΦΣΥ. Τα στάδια της δημιουργίας αυτού του ταμείου ήταν καταρχάς ε, βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που βοήθησε και μας βοήθησε να έχουμε χρηματοδότηση της τάξης των 20 εκατομμύριων ευρώ για το ταμείο αυτό, το CAP3 RI και τον Οκτώβριο του 2015 στα μέσα Οκτωβρίου, κάποιους μήνες λοιπόν μετά από την, ένταξη, την έναρξη, ε, θεωρηθήκαμε διαχειριστής ε, του Ταμείου αποφασίστηκε ότι θα υπάρχει και συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με 15 εκατομμύρια ευρώ και το Νοέμβριο του 2015 συστήθηκε το Ταμείο. Έχουμε λοιπόν ε, ε, κεφάλαιο το οποίο μπορούσαμε να επενδύσουμε και εμείς, 12,5 εκατομμύρια και 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τεχνική βοήθεια. Τα πάντα προχώρησαν πάρα πολύ γρήγορα. Τον Ιούλιο του 2015 μέχρι τον Νοέμβριο του 2015, δηλαδή τέσσερις μήνες, καταφέραμε να τα κάνουμε όλα και από τον Νοέμβριο του 2015 συστήθηκε το Ταμείο. Σήμερα έχουμε την εικόνα του Ταμείου, έχουμε 12,5 εκατομμύρια από τα 12,5 του Ταμείου Περιφερειακής Ανέπτυξης τα οποία επενδύθηκαν, έχουμε την Κρεντή Αγκρικόλ που επένδυσε κάποιο ποσό και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που ε, χρηματοδότησε περίπου με 20 εκατομμύρια ευρώ. 8 εκατομμύρια είχαμε από την Κρεντή Αγκρικόλ και επομένως βλέπετε ότι έχουμε τέσσερις πρωταγωνιστές και έχουμε και την ομάδα ε, North Capital η οποία ε, συμμετέχει εδώ και τρεις μήνες και έχει ε, προσφέρει 3 εκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλούς ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι έρχονται να μας δουν για να δουν αν μπορούν να επενδύσουν χρήματα στο ταμείο. Υπήρχε, για παράδειγμα, μια εταιρεία που ήθελε να ε, επενδύσει 6 εκατομμύρια ευρώ. Το σκεπτικό μας βέβαια δεν είναι να πάρουμε αυτά τα χρήματα, αλλά καταρχάς να τα επενδύσουμε. Τώρα, σχηματικά, έχουμε κάτι αντίστοιχο με προηγουμένως και εδώ στην ίδια διαφάνεια βλέπουμε ότι ε, έχουμε και κάποια πράγματα όσον αφορά τις επενδύσεις μας. Το CAP 3 αρι διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή 40,5 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε επενδύσεις και από επιχειρήσεις και έχουμε και κάποιες ε, εκτιμήσεις και φτάνουμε περίπου στα 200 ε, εκατομμύρια ευρώ. Το πενταπλάσιο δηλαδή. Στις τράπεζες σκεφτείτε τι γίνεται. Στόχοι του Ταμείου και σε αυτό άλλωστε θα κρυθούμε, είναι καταρχάς να προσπαθήσουμε να έχουμε μια οικονομία η οποία βασίζεται σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, ε, να μειώσουμε κατά τέσσερα ε, τις κατά ένα συντελεστή 4 τις εκπομπές του αερίου του θερμοκηπίου και να είμαστε 60% πιο αποτελεσματικοί. Οι διάφορες προτεραιότητες επενδύσεων του Ταμείου βασίζονται στην ενεργειακή μετάβαση ε, για τους τέσσερις βασικούς πυλώνες και στην κυκλική οικονομία για, τους, ε, για τον τελευταίο πυλώνα. Στη, ε, θέλουμε να έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή ηλιακή ενέργεια. είναι περίπλοκο βέβαια σε όλες τις περιοχές της Γαλλίας. Βιομάζα. Στη συνέχεια έχουμε και ό,τι έχει σχέση με τη διαχείριση της ενέργειας, το, e, τα ή e e, δίκτυα, έξυπνα δίκτυα ενεργειακή απόδοση, ευφυή κινητικότητα, οτιδήποτε είναι οικολογικό και φυσικά και την κυκλική οικονομία που είναι ε, η κατάλληλη διαχείριση αποβλήτων ε, και για τις βιομηχανίες αλλά και ε, για διάφορες κοινότητες. Τα κριτήρια επενδύσεων μα δείχνουν ότι πρόκειται καταρχάς για ένα σχέδιο το οποίο έχει σχέση με την τρίτη βιομηχανική επανάσταση ε, θέλουμε ένα κεφάλαιο ανάπτυξης βεβαίως για τις επενδύσεις. Δεν ξέρω αν είστε και εξοικειωμένοι με τα ταμεία επενδύσεων ε, αυτή τη μορφή. Αυτό σημαίνει επενδύουμε συνήθω σε όρμες επιχειρήσει, έχουν κάποιο κύκλο εργασιών ε, και έχουν και κάποιο ποσοστό εξαγωγών και χρειάζονται χρηματοδότηση και ενίσχυση του ιδίων κεφαλαίων για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Όπως σας είπα προηγουμένως, εμείς επενδύουμε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε κάποια προγράμματα, αλλά σε σχέση αυτό με τις διάφορες περιφέρειες της Γαλλίας και υπάρχουν και κάποια προγράμματα τα οποία έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης για την περιοχή. Προσπαθούμε να δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά του Ταμείου. Σήμερα λοιπόν θεωρούμε ότι είμαστε μέτοχος με μειοψηφικό κεφάλαιο. Δηλαδή, επενδύουμε και παίρνουμε λιγότερο από το 5% των ε, ε, μεριδίων της εταιρείας. Αυτό συνήθως είναι 15 με 20%. Εμείς επενδύουμε μεσοπρόθεσμα, λίγο πολύ, ε, αναφερόμαστε στα κονδύλια της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης. Ε, πρόκειται λοιπόν για μια επιχείρηση που κάνει επενδύσεις δεν θα έχουμε απεριόριστη διάρκεια. Ο στόχος είναι να αποδώσουμε τα χρήματα στους επενδυτές από το 2027. Δηλαδή σε 7 χρόνια έχουμε ένα ορίζοντα 7 ετών. Ε, ε, το μέγεθο των επενδύσεών μας είναι τη τάξη του 1 εκατομμυρίου ευρώ τουλάχιστον, που σημαίνει ότι μπορούμε να περιορίσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, τα έργα στα οποία μπορούμε να επενδύσουμε. Η τρίτη βιομηχανική επανάσταση είναι επανάσταση, λοιπόν είναι κάτι καινούριο και χρειαζόμαστε πάρα πολλέ μικρομεσαίε, ε, μάλλον συγγνώμη, έρχονται να μα δουν πολλέ επιχειρήσει. Εμείς βέβαια έχουμε το σκεπτικό ότι δεν μπορούμε απαραίτητο να επενδύσουμε σήμερα. Βοηθάμε να αναπτυχθούν αυτά τα προγράμματα μέσω ενδιαμέσων από άλλα ταμεία τη περιοχή. Εάν λοιπόν χρειάζονται απαραίτητα ταμεία, του φέρνουμε σε επαφή με ιδιώτες επενδυτές εκτός του δικού μας του προγράμματος δίνεται συνήθις χρηματοδότηση, ε, είτε με μερίδια είτε με ε, μετατρέψιμα ομόλογα και ε, προσφέρεται και τεχνική ε, βοήθεια. Μπορούμε να επενδύσουμε μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της επένδυσης. Αυτό φυσικά με συμμετοχή και άλλων επενδυτών. Υπάρχει ένα ποσό το οποίο μπορούμε να δώσουμε λοιπόν αρχικά στην επιχείρηση, το οποίο ε, ε, υποχρεωτικά όμως θα πάει προς την cap ε, 3RI. Αν μας πει κάποιος ότι χρειαζόμαστε 10 εκατομμύρια ευρώ, τα τρία θα τα δώσουμε εμείς και τα λεφτά θα τα δώσουν είτε ιδιώτες επενδυτές, είτε θα τους βρούμε άλλους επενδυτές κλπ. Και κυρίως μας ενδιαφέρει και η τεχνική συνδρομή. Έχουμε 2,5 εκατομμύρια τεχνική συνδρομής. Αυτά τα 2,5 εκατομμύρια που είναι από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι τελείως διαφορετικά για μας. Δηλαδή, ε, έχουμε ένα περιφερειακό ταμείο επενδύσεων και θέλουμε να έχουμε και ένα εξειδικευμένο ταμείο επενδύσεων που είναι εξειδικευμένο σε ενεργειακά θέματα. Πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σπάνιο στην ευρωπαϊκή αγορά, μπορεί και να είναι μοναδικό και μας επιτρέψει ε, να έχουμε μεγαλύτερη εξειδίκευση ε, για τα ταμεία επενδύσεων και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις στις οποίες θέλουμε να επενδύσουμε χάρη σε αυτό το χαρτοφυλάκιο ε, ενισχύσεων των 2,5 εκατομμυρίων. Έχουμε άμεση διαχείριση και μπορούμε να επενδύσουμε μέχρι και 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση και ανά έργο. Άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνική συνδρομή νωρίτερα για να μπορέσουμε να επενδύσουμε στη συνέχεια στην επιχείρηση. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι επενδύουμε και μετά θα σας δώσουμε άλλες 100.000 ευρώ για να αυξήσουμε το ποσό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να γίνει πριν ε, γίνει η αρχική επένδυση. Και ε, οι επιχειρήσει αυτές μας προτείνουν κάποιο έργο στο οποίο δυνητικά θα μπορούσαμε να επενδύσουμε αλλά όχι υποχρεωτικά. Ε, Και βλέπετε τώρα ότι υπάρχουν δύο σημεία τα οποία μας ενδιαφέρουν. Καταρχάς έχουμε στήριξη, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε λοιπόν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν τα προγράμματά τους. Έχουμε περίπου 200.000 ε, ευρώ έχουν δοθεί για να επενδύσουμε σε αυτά τα τις επιχειρήσεις και έχουμε και την αξιολόγηση, στην οποία βλέπουμε μέχρι ποιο σημείου η επιχείρηση θα μπορέσει να έχει και κάποιον αντίκτυπο για την τρίτη βιομηχανική επανάσταση και την οικονομία. Ε, να δούμε δηλαδή κατά πόσον όλα αυτά θα γίνουν ε, σε σχέση με άλλα θέματα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, ε, τι συνέπειες υπάρχουν για εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κλπ. Η γενική στόχη λοιπόν του Ταμείου μας είναι να είμαστε παράγων επενδυτικών κεφαλαίων που ε, θα έχουμε και διάρκεια στο χρόνο και θα υπάρχει και διαχείριση, θα βοηθούμε ε, τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Μακροπρόθεσμα είμαστε μια εταιρεία επενδύσεων, μπορούμε να μείνουμε λίγο παραπάνω από ότι μια κλασική επενδυτική εταιρεία και χρειαζόμαστε φυσικά και συμμετοχή του τοπικού κλάδου. Να σας πούμε λίγο τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ε, σας είπαμε ότι συσταθήκαμε στις, το Δεκέμβριο του 2015. Το Ταμείο ξεκίνησε ε, καταρχάς και θέλαμε να συστήσουμε τα πάντα, να βρούμε και την ομάδα μας. Έχουμε 110 προγράμματα τα οποία είχαν σχέση με την τρίτη βιομηχανική επανάσταση και την περιοχή της Γαλλίας. Ε, αναλύσαμε τις λεπτομέρειες σε 45 προγράμματα. Έχουμε προχωρήσει και έχουμε ε, υποστηρίξει 7 επιχειρήσεις τις οποίες ε, παρουσιάσαμε και στην Συμβουλευτική Επιτροπή Επενδύσεων η οποία αποτελείται από εμπειρογνώμονες ε, και μετόχους και από τα 7 τα οποία παρουσιάστηκαν τελικά έγιναν δύο επενδύσεις. Η συμφωνία έγινε με το Συμβουλευτική Εταιρεία. Ε, το πρώτο με την Τρεκάν και το δεύτερο με την Αστραντέκ. Οι επενδύσεις αυτές ξεκίνησαν ε, για το 2015 με μια εταιρεία που λέγεται DREKAN που είναι στην, ε, ε στις ηλεκτρικές τουρμπίνες. Ε, ασχολούνται με την επισκευή ηλεκτρικών συσκευών που έχουν τουρμπίνες. Πώς μπορούμε να επισκευάσουμε ένα κινητήρα ε, και από εκεί και πέρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, τους κινητήρες αυτές. Έχουμε λοιπόν κυκλική οικονομία εδώ πέρα και πρόκειται για μια εταιρεία η οποία ε, έχει διάφορες περιοχές στη Γαλλία και θέλει να αναπτύξει ένα πρόγραμμα στις διάφορες περιφέρειες της Γαλλίας. σε 15 χρόνια θα πρέπει να αλλάξει ή να ε, σταματήσει ε, και έχουμε εδώ αυτές τις αιωλικές τουρμπίνες τις οποίες χρησιμοποιούν. Θα δημιουργήσει και θέσει εργασία, γιατί θα υπάρξει μια θηγατρική και ελπίζουμε να έχουμε 60 θέσεις εργασίας σε 5 χρόνια σε συγκεκριμένη περιοχή της Γαλλίας και έχουμε περίπου 10 εκατομμύρια επενδύσεων για να μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε επιπλέον εγκαταστάσεις οι οποίες θα σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες. Όλα αυτά ε, από μία επένδυση 1,5 εκατομμυρίου. Δηλαδή έχουμε όντως το πενταπλάσιο της επένδυσης ε, ε, όσον αφορά το επενδυτικό κεφάλαιο. Η δεύτερη επιχείρηση στην οποία επενδύσαμε πρόκειται για μια νέα επιχείρηση, λέγεται Astradec μια επιχείρηση η οποία κάνει συλλογή απορριμμάτων και ανακύκλωση και ασχολείται με την ανακύκλωση και την αξιοποίηση αποβλήτων. Ε, έχει κάποια προγράμματα τα οποία είναι πάρα πολύ καλά για την τοπική οικονομία και αναπτύσσεται πάρα πολύ ε, μέσω και εξωτερικής βοήθειας. Σήμερα, δεν ξέρω αν τα βλέπετε καλά, σας μίλησα για 7 προγράμματα τα οποία παρουσιάστηκαν στο ε, συμβουλευτικό όργανο. Έχουμε λοιπόν δύο τα οποία έχουμε ε, ήδη υλοποιήσει και έχουμε άλλα πέντε και τα οποία θεωρούμε ότι είναι εμβληματικά ε, χαρακτήρα. Ένα αφορά την κυκλική οικονομία, μέταλλο και ενέργεια και το άλλο ένα πρόγραμμα για την ανάκτηση της θερμότητας την οποία θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε κύκλους βιομηχανικής θερμότητας στη συνέχεια. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή, τα οποία μπορούμε να τα δούμε σε σχέση με τα διάφορα προγράμματα που αναπτύσσουμε, χάρη στη βοήθεια και των επενδυτών. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Ah, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βατρή. Νομίζω ότι όσοι παρακολούθησαν ε, με προσοχή τις ε, ομιλίες και τις συγκεκριμένη ομιλίες στο τέλος. Ε, έχουν μάθει τα πάντα για την 4-3 ri Είναι σαν να πρόκειται για ένα μικρό περιφερειακό εύση με προσανατολισμό την τρίτη βιομηχανική επανάσταση. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν ο σκοπός ε, της επιλογής, αλλά νομίζω ότι συνάδει αρκετά με μια περιφερειακή προσαρμογή του ευρωπαϊκού αυτομοντέλου. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους ε, ευρωβουλευτές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ήδη ο κύριος Όλμπιχτ πήρε το λόγο, ο κύριος Μάνκα. Τώρα ο κύριος Φερνάντες είχε συζητήσει από πριν το λόγο. Το σημειώνω. Λοιπόν, ο κύριος Φερνάντες, ο εισηγητή μας. Ευχαριστώ. Θα είμαι εξαιρετικά λακωνικός. Ο σκοπός του ΕΦΣΙ είναι να λειτουργεί επιπρόσθετα. Δεν μπορεί να πάρει μόνο τα προγράμματα πολύ υψηλού ρίσκου, αλλά σίγουρα παίρνει τα υψηλού ρίσκου. Γιατί αν δεν είναι υψηλού ρίσκου, τότε δεν ε, έχει αυτή την προσθετική δράση. Πρέπει να κάνουμε αυτό το blending, ε, αυτή την διασύνδεση με το Ταμείο ε, Συνοχής μετά την ε, παρακολούθηση του Γιον, συγγνώμη, την παρέμβαση του Γιάννη Όλμπριχτ ε, είναι κάτι που πρέπει να θίξουμε. Τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τι συμφωνίε σχέσεις, σχέση, έχουν ήδη τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ε, τέτοια χρηματοδοτικά μέσα, επενδυτικά ταμεία. Υπάρχει κάτι το οποίο θα ήταν ίσως αρνητικό, να κάνουμε ένα συνδυασμό αλλά τώρα, να παίρνουμε χρήματα, κονδύλια από την πολιτική συνοχής για να τα διοχετεύσουμε στο ΕΦΣΥ θεωρώ ότι όχι δεν είναι σωστό. Γιατί αυτό δίνει έτσι τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να έχει μια ιδιαίτερα διακριτική στάση και να πει όχι, δεν χρησιμοποιεί τα ταμεία όπω θα έπρεπε. Πρέπει αυτά τα κονδύλια να τα πάρει από την πολιτική συνοχή, για παράδειγμα, για να τα βάλει σε ένα χρηματοδοτικό μέσο, αν θέλει να υιοθετηθεί το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν ε, περί αυτού πρόκειται. Εάν όμως είναι έτσι, τότε πιστεύω ότι θα ήταν μια πολύ κακή ιδέα. Αν μιλούμε για έναν βαθμό ευελιξίας και έτσι να πούν κάποια κρατημέλη ότι εγώ τώρα ε, χρειάζομαι να ενισχύσω τον μηχανισμό περιφερειακής ή εθνικής χρηματοδότησης. Εκεί θα έλεγα μάλλον ναι. Και αυτό θα εξαρτάται από τη βούληση του κράτους μέλους. Δεν θα ήταν δηλαδή κάτι που θα επιβαλόταν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή από την διαχείριση του ΕΦΣΥ. Επομένω, η συμπληρωματικότητα είναι που έχει σημασία εδώ για να διαμορφώσουμε συνέργειες με το ΕΦΣΥ ή άλλων χρηματοδοτικών ε, ε, μέσων με τα θετικά ταμεία. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό σκέλος. Όμως, το θέμα είναι περί τίνος πρόκειται. Εάν μιλούμε για τη δυνατότητα άντληση κονδυλίων από την πολιτική συνοχή για να τα διοχετεύσουμε στο ΕΦΣΥ ή ότι το ΕΦΣΥ θα μας λέει πώς ε, θα δαπανίσουμε τα κονδύλια που έχουμε στην πολιτική συνοχή, νομίζω ότι αυτό δεν θα πρέπει να το δεχθούμε. Ένα άλλο ερώτημα τώρα. Για ποιο λόγο έχουμε κακή εκτέλεση των κονδυλίων των ιδιωτικών ταμείων αυτή τη στιγμή είναι ο κανόνα 1 3 που λέμε συχνά, λέει συχνά μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε μιλούμε για την απλούστευση. Όταν μιλάμε μάλλον για απλούστευση, εγώ είμαι λίγο διστακτικό γιατί σε κάθε πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο το ίδιο πράγμα λέμε για απλούστευση και τελικά τα περιπλέκουμε τα πράγματα. Ποια είναι λοιπόν η απλούστευση που πρέπει να επιτύχουμε αυτή τη στιγμή ταχύτατα για να βελτιώσουμε αυτή την κακή εκτέλεση που έχουμε αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τα διευθυντικά ταμεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Κέρμιλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ομιλητές μας ε, για τις ε, πολύ διαφοροποιημένες μεταξύ τους ε, ομιλίες, οι οποίες πραγματικά απέφυσαν και πολύ συμπληρωματικές. Αυτή η διαφορετικότητα, αν θέλετε, τονίστηκε για μία ακόμα φορά σε αυτές τις παρεμβάσεις και νομίζω πως εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. δηλαδή νομίζω πως αυτό που υπόθηκε πολύ εύστοχα από ένα από τους ομιλητές είναι να λέμε ότι όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να προβλέπονται με πολύ αυστηρό τρόπο, έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες αρχές ελέγχων και ούτω καθεξής και από την άλλη πλευρά να λέμε ότι θέλουμε ένα προϋπολογισμό ο οποίος θα ε, προσανατολίζεται στις επιδόσεις, τον οποίο θα ελέγχω και αυτό στη συνέχεια. Δηλαδή, εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να επανεξετάσουμε τι υφιστάμενε διαδικασίε και όπου αυτό χρειάζεται να τι καταργήσουμε. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, με του νέου κανόνε, ουσιαστικά θα έχουμε μία ε, διπλή διαδικασία, διπλέ διαδικασίε, ε, με αποτέλεσμα βέβαια, τελικό αποτέλεσμα, χαμηλότερη ποιότητα ε, στην εκτέλεση του προπολογισμού και όχι υψηλότερη ποιότητα. Και θα πρέπει βέβαια να λαμβάνουμε υπόψη μα και το τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, εάν κάποιος ε, θεωρεί ε, πως εάν αναλάβει υπερβολικές ευθύνες ή κινδύνους, ε, ενδεχομένως τα πράγματα να αποβούν, να έχουν άσχημη εξέλιξη, φυσικά δεν θα είναι διατεθειμένο το λόγο άτομο να προβεί σε τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις. Εάν θέλουμε λοιπόν να μην ε, προβούμε σε βαθιέ τομέ, τότε ουσιαστικά θα κάνουμε μικροπαρεμβάσει με αποτέλεσμα να αυξάνουμε όλο ένα και περισσότερο την περιπλοκότητα και την γραφειοκρατία. Νομίζω λοιπόν πω εάν θέλουμε να συζητήσουμε για αποτέλεσμα, τότε θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλουμε στην υψηλότερο, στο υψηλότερο, στο καλύτερο αποτέλεσμα και πώ μπορούμε να ε, εμπιστευτούμε εδώ τα κράτη-μέλη, στο βαθμό δηλαδή που αυτό είναι δυνατό. Ε, όπου δηλαδή τα κράτη-μέλη μπορούν να αναλάβουν μόνα τους ε, το τμήμα της εκτέλεσης, ε, γιατί θα πρέπει να εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε πάρα πολύ στη μείωση του διοικητικού άκθους. Και από εκεί και μετά να πω ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι χρηματοδότηση ενό προπολογισμού. Υπάρχουν δηλαδή άμεσε επενδύσει, υπάρχουν πάνε, υπάρχουν και εγγυήσει, οι οποίε χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίε, αλλά όλο ένα και περισσότερα ε, περιπλέκουμε και σε σχέση με αυτές τις ε, πηγές αν θέλετε και τις, ε, του, του δηλαδή τα νέα εργαλεία, τους νέους μηχανισμούς που δημιουργούμε. Γιατί δηλαδή ή τι μας αποδεικνύει ότι όσα χρηματοδοτούμε αυτή τη στιγμή μέσω του ΕΦΣΥ δεν ήταν δυνατό να χρηματοδοτηθούν μέσω της Τράπεζας Επενδύσεων. Δεν μπορούσε δηλαδή να δώσει εγγυήσεις για όλα αυτά τα project ήδη η Τράπεζα Επενδύσεων. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο θα πρέπει ε, τα κονδύλια τα οποία ε, ε, θέτουμε στη διάθεση για αξιοποίηση θα πρέπει να δούμε κατά πόσο έχουμε τόσο έχουμε δώσει τόσο μεγάλη έμφαση στη συμπληρωματικότητα, γιατί ακούσαμε και από όλε τι παρεμβάσει ότι τελικά κανένα δεν εντόπισε κάπου μία πραγματική συμπληρωματικότητα μεταξύ των εργαλείων που δημιουργούμε. Δηλαδή, ναι, θα πρέπει να ε, ε, κάνουμε κάποιε ρηξικέλευτε ε, λύσει εδώ, να εφαρμόσουμε κάποιε ρηξικέλευτε λύσει, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και το τι σημαίνει με τα πελαιότερα εργαλεία, αλλιώ δεν θα κάνουμε τίποτα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μανατίτσα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ όλους τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους και Λυπούμε που έλειψα για περίπου 15 λεπτά για μια ψηφοφορία και δεν άκουσα ε, την ε, τσεχική παρουσίαση. Είδα όμως τις διαφάνειες. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Νόνες Φερέρ ότι έχουμε έναν τόσο περίπλοκο προπολογισμό που τελικά δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε τα απλά και πολύ βασικά ερωτήματα. Τι θέλουμε να πετύχουμε, τι έχουμε πετύχει και αν θέλουμε να υπάρξει η διασύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκού Προπολογισμού και Ευρωπαϊκής Στρατηγικής δεν είναι εύκολο να το πετύχουμε. Έχουμε ένα στρατηγικό έγγραφο το 2020, τώρα πρέπει να προετοιμάσουμε το καινούργιο και το 2030. Χρειαζόμαστε λοιπόν σαφείς συνδέσεις με τον προπολογισμό. και να δούμε τι κάνουμε αυτή τη στιγμή στο προπολογισμό μας για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε στο στρατηγικό μας έγγραφο. Δεν είναι βέβαια απλό εγχείρημα αυτό. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να ε, τροποποιήσουμε τον προπολογισμό, να τον απλουστεύσουμε. Και αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως, πρέπει να δώσουμε έμφαση στα έργα. οι τελικοί δικαιούχοι και όσοι υλοποιούν τα προγράμματα να μπορούν εύκολα ε, να διευθετήσουν όλες τις διαδικασίες ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, απευθυνόμαστε σε ένα σημείο επαφή, σε ένα όργανο που μας δίνει κάποια απάντηση. Και απέχουμε πάρα πολύ από αυτό το σημείο, γιατί ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να μας απαντήσει τι χρηματοδοτείται από ποιον. Γιατί έχουμε τόσες διαφορετικές πηγές ε, για τα ίδια πράγματα. Στην παρουσίασή σας ε, μας μιλήσατε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά το ίδιο ισχύει και για τις πόλεις, ε, για τους φορείς καινοτομίας, για, για οποιονδήποτε άλλο. Επομένω, είναι εξαιρετικά σύνθετη η κατάσταση και για όσους υλοποιούν τα προγράμματα και για όσους πρέπει κάτι να κάνουν για να έχουν ε, τα επιτεύγματα που επιθυμούν. Αν λοιπόν δεν αλλάξουν τα πράγματα στο μέλλον, ε, θα είμαστε ακόμα πιο μακριά από την πραγματικότητα και από τους πολίτες μας και αυτό πρέπει να αλλάξει. Γιατί πρέπει πραγματικά να είμαστε πολύ κοντά στο πολίτη, ε, με μια πρακτική και ρεαλιστική διάθεση, να βρούμε πρακτικές λύσεις. Και εδώ συμφωνώ πολύ τους μαζί σας. Πρέπει να ξεκινήσουμε μία ιδιαίτερα ε, αναλυτική συζήτηση σε αυτό το σημείο. Κάτι άλλο τώρα συνεχώς προσπαθούμε να σβήσουμε πυρκαγιέ με τον προπολογισμό, δρούμε πυροσβεστικά και τελικά έχουμε τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, το Ταμείο ε, Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Αλλά τελικά ε, απλώς προσπαθούμε να αντιδράσουμε στην οικονομική κρίση. Έτσι πρέπει να είναι ο Ευρωπαϊκός προπολογισμό είναι σαν μια κυβερνητική παρέμβαση κατόπιν ε, εξαιτία μάλλον μιας οικονομική κρίσης. Η τελευταία συζήτηση που κάναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πώς θα αξιοποιήσουμε την πολιτική συνοχή για τους σεισμούς. Εντάξει, σαφώ και θα αναγκαστούμε να δράσουμε και περιοριστικά, αλλά ο προπολογισμό είναι το κατάλληλο μέσο για να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα. Εγώ νομίζω ότι ακολουθούμε λανθασμένη κατεύθυνση και γι' αυτό είμαστε διστακτικοί όταν μιλούμε για ε, συνδυασμό των, του ΕΦΣΙ και των διαφορετικών κυβερνητικών ταμείων, γιατί δεν βλέπουμε κάποιο νόημα πια. Στην αρχή όταν υιοθετήθηκε το ΕΦΣΥ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα ε, το παρουσίασε, μα είπαν ότι θα αφορούσε μόνο ιδιωτικέ επενδύσει σε υψηλού ρίσκου προγράμματα και τώρα ξαφνικά το συνδυάζουμε με την πολιτική συνοχή. Εδώ φτάσαμε. Δεν καταλαβαίνω πια τον προπολογισμό και είμαι η Δήμων στα ζητήματα ε, του προπολογισμού γιατί στην Κροατία ήμουν στο Υπουργείο Οικονομικών για 15 χρόνια και ασχολούμουν με τα θέματα του προπολογισμού και την πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ. Κανονικά οι βιογνώμονες μας ε, πρέπει να μας ε, ε, βοηθήσουν να ξαναβρούμε τον ίσιο δρόμο. Ο κύριος Βανίστελρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Άκουσα ένα τμήμα της και έχω και τι διαφάνειε. Εγώ είμαι Ολλανδός και είμαι θετικά διακείμενος γιατί έχουμε και ανεπτυγμένη αίσθηση του σχεδιασμού και της ε, βιομηχανοποιημένης συνεργασίας της ε, περιφέρειας μας, όπως και η Βόρεια Γαλλία. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με αυτά τα πράγματα, αλλά αν πάτε στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και σε άλλες περιφέρειες, δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες απαιτήσει. Και εφόσον ε, βασιζόμαστε πολύ στην στην πλευρά της ζήτησης, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια σαφή εικόνα της Ευρώπης. Γιατί η εδαφική διάσταση είναι εξαιρετικά σημαντική. Δεν είναι το εύση βάζει το κερσάκι στην τούρτα δεξιά και αριστερά χωρίς καμία σύνδεση. Στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στις περιφέρειες, ε, στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό ικανότητας, γιατί πρέπει να υπάρχει και εμπειρογνωμοσύνη σε αυτού τους κλάδους. Νέα βιομηχανική επανάσταση χωρίς ε, ανθρώπους δεν μπορούμε να έχουμε. Επομένω, χρειαζόμαστε έναν ολοκληρωμένο οριζόντιο προγραμματισμό στι πόλει και στι περιφέρειε που αποτελούν τη βάση για αυτή τη νέα δημιουργία πλούτου. Ήμουν σκιώδης ε, σε αυτή την ιστορία με την πρόταση Omnibus ένα από τα στοιχεία που είπαμε σήμερα το πρωί, στα οποία είπαμε όχι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι απαραίτητο να παίρνουμε χρήματα από τους ε, φακέλους των κρατών μελών πίσω στην ΕΤΕΠ. Να δείχνουμε εμπιστοσύνη στα κρατημέλη και να δώσουμε στα κρατημέλη δυνατότητα, όπου αυτό είναι δυνατόν και απαραίτητο, να αξιοποιήσουν αυτούς τους μηχανισμούς ε, υψηλού ρίσκου είτε ε, με την ε, υποδοχή ιδιωτικών κεφαλαίων είτε με επιδοτήσεις. για πολλές κατηγορίες μακροχρόνιων, μακροπρόθεσμων, υψηλού, ρίσκου επενδύσεις δεν γίνεται αυτό. Να, δώσουμε, λοιπόν, να δείξουμε την εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη και μετά τα κράτη-μέλη μαζί με τα υπόλοιπα επίπεδα, σε διαφορετικά μέρη που είναι συνεπενδυτέ και συνδιαμορφωτέ της πολιτικής να δουν σε ποιο βαθμό θα αξιοποιήσουν αυτά τα, αυτούς τους μηχανισμούς ε, τύπου εύση. Δεν χρειάζεται κάθε χώρα να το αξιοποιεί το FC. Όχι. Και μετά. Πρέπει να σταματήσει επιτέλους αυτή η συζήτηση για το blending, για την ανάμειξη διαφορετικών στοιχείων. Μα γιατί μιλάμε. Υπάρχουν στόχοι στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη και για την ε, πολιτική συνοχή. Και το FC μπορεί να βοηθήσει σε κάποια στοιχεία, αλλά το blending είναι τρελό. Κάποιες φορές χρειαζόμαστε 10 ε, χρόνια ε, για να ευοδοθεί μια προσπάθεια. Το ακούσαμε και από τη βιομηχανία προηγουμένως. Περιφερειακή διάσταση, χρονική διάσταση και η πολυμορφία στην Ευρώπη. Αν προσπαθήσουμε όλοι να τα κάνουμε απλά και εύκολα, δεν γίνεται. Και δεν πρέπει να φτάσουμε σε μια κατάσταση που να θεωρούμε ότι όλη η Ευρώπη είναι ίδια, γιατί δεν ισχύει. Κάποιες χώρες είναι πιο προηγμένες. Ήδη ακολουθούν αυτή την πολιτική. Δεν χρειάζονται το εύση. Στην Ολλανδία δεν χρειαζόμαστε το εύση. Αλλά εφόσον έχει δημιουργηθεί το χρησιμοποιούμε. Αλλά και η αγορά από μόνη της μπορεί να το κάνει χωρίς ε, το εύση. Εύκολα. Αλλά τέλος πάντων δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε την ίδια μεθοδολογία στη συσκελία. Γιατί τελικά δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Εσεί είπατε στόχοι για το 2050. Αχ, πόσο χαίρομαι όταν το ακούω αυτό. Θέλουμε μακροπρόθεσμο όρεμα και η κάθε χώρα να συμμετάσχει όπως επιθυμεί. Αν κάποιο θέλει να ανταποκριθεί στην έκκλησή μου, βεβαίω με τα χαρά να τον ακούσω. Ε, ε, Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και για την έκκλησή σας. Ίσως κάποιος θέλει ε, να πάρει το λόγο ο κύριος Μάνκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν ανοίξετε μια ματιά στα προγράμματα του ΕΦΣΥ, διαπιστώσετε ότι για παράδειγμα ένα κράτος μέλος ε, το οποίο ήθελε να κατασκευάσει έναν αυτοκινητόδρομο έπρεπε να αυτοχρηματοδοτήσει το 95% και να λάβει ε, συμπληρωματικά 5% από το ΕΦΣΙ. Έχουμε δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες έχουν συμβεί για παράδειγμα και στη Γαλλία ή αλλού όπου υπάρχουν project τα οποία χρηματοδοτούνται αλλά τα οποία θα μπορούσαν ούτως ή άλλως να υλοποιηθούν ε, με αμυγός σε κρατική χρηματοδότηση. Οπότε δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις δεν ξέρω αν πραγματικά ήταν απαραίτητη η συνεισφορά από την πλευρά του ΕΦΣΥ. Όταν κάνετε λόγο για αυτό το blending, εντάξει, πράγματι έχουμε προτείνει μια αποσυρά ε, νέων μεθόδων και στο πλαίσιο του, της πρότασης Omnibus ε, και πράγματι δεν είναι δυνατόν για όλα τα κράτη-μέλη να αξιοποιούν όλα τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο των ε, ΕΔΕΤ οπότε εκείνα τα μη αξιοποιούμενα κονδύλια θα πρέπει να διασφαλίσουμε να αξιοποιούνται καλύτερα σήμερα. Ήδη το κάνουμε σε κάποιο βαθμό σήμερα αλλά θα πρέπει όπω είπε και ο συνάδελφο Μανίστερο, το κάτω μέλο το οποίο δεν απορροφά αυτά τα κονδύλια να αποφασίζει τι μπορεί να κάνει περαιτέρω με αυτά, πώ μπορεί δηλαδή να τα αξιοποιήσει περαιτέρω. Και νομίζω πω ε, για το FC20, τη νέα δηλαδή έκδοση του, θα πρέπει να σκεφτούμε ακριβώ τέτοιε λύσει. Πώ δηλαδή θα είναι δυνατόν να αξιοποιείται περαιτέρω αυτή η χρηματοδότηση. Όταν πρωτοδημιουργήθηκε το FC, ο σκοπό μα ήταν να αξιοποιείται μόνο σε περιπτώσει εκείνε ε, έργων Λοιπόν τα οποία δεν θα ήταν δυνατόν να υλοποιηθούν χωρίς τη χρηματοδότησή του. Δεν ε, είναι λοιπόν θεμητό το ότι βλέπουμε τώρα να χρηματοδοτούνται έργα τα οποία θα μπορούσαν ούτως ή άλλως να υλοποιηθούν, χωρίς δηλαδή ε, το ΕΦΣΙ. Συμφωνώ επίσης με αυτό που υπόθηκε ότι θα πρέπει ε, κάποια στιγμή να δημιουργηθούν και ενιαίες διαδικασίες ελέγχου, κοινό δηλαδή έλεγχος, ε, και ίσω θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πιστοποιημένο οργανισμό ελέγχων ο οποίο θα προβαίνει για παράδειγμα σε έναν ενιαίο έλεγχο για κάθε έργο. Παρ' όλα αυτά βέβαια η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ύπαρξη αμφιβολιών να προβαίνει σε ε, συμπληρωματικού ελέγχου εφόσον τους θεωρεί απαραίτητου. Αυτά από την πλευρά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα έχει ο Γιάνν Ολμπριχτ. Παρακαλώ. Ναι. Συμφωνώ με τον ε, συνάδελφο που μίλησε προηγουμένως και είπε ότι έχουμε τη δυνατότητα να ε, θίξουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα το οποίο δεν ακολουθεί την πεπατημένη. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία πρέπει να συζητήσουμε μέσα στις επόμενες ημέρες και μήνες. Πρέπει να συζητήσουμε το νέο ΠΔΠ και νέα στοιχεία της ε, πολιτικής συνοχής. Υπάρχουν στοιχεία χρήσιμα για αυτή τη συζήτηση. Πρώτον, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς ε, να δείχνουμε πιστοσύνη ένα στον άλλον και προς τα κρατημέλη και προς τους τελικούς δικαιούχους. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, πρέπει να απλουστεύσουμε τη διαδικασία και μετά να ελέγξουμε. Αλλά με ένα πολύ απλό τρόπο. Χωρίς την εμπιστοσύνη δεν θα πάμε πουθενά. πολύ συχνά λέμε ότι θέλουμε και την πιταλόκληρη και το σκύλο χορτάτων. Επομένω, το πρόβλημα είναι ο προπολογισμό. Ε, είναι αυτό ακριβώ αυτό που έχουμε, παρακολου... Ε, που έχουμε ήδη εντοπίσει. Δεν είναι λοιπόν, ο μήπως ο προπολογισμό βάσει επιδόσεων είναι απλώς ένα μότο. Είναι μια πραγματική τεχνική πρόταση. Γιατί τότε υπάρχει πρόβλημα. Είναι αυτό που είπε ο Λάμπερτ στο τέλο. Είμαστε υπέρ τη συμπληρωματικότητα των συνεργειών, σίγουρα, τη ολοκληρωμένη προσέγγιση, αλλά με σοβαρό τρόπο. Είμαστε κατά όμω του blending. Γιατί έτσι, αν τα μπλέξουμε όλα, θα πέσουμε στην παγίδα και τελικά ε, οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν σε πολλές γενικές ευθύνσεις και να υποστούν έλεγχο από όλους. Όταν εξετάζουμε το Omnibus, ε, δεν είναι ότι δεν θέλουμε τη διασύνδεση με το ΕΦΣΥ, αλλά το Omnibus έχει ως ειδικό στόχο, στόχο να απλουστεύσει τις διαδικασίες από αυτή την άποψη. Είναι για τώρα λοιπόν η πρόταση Omnibus. Χρειαζόμαστε ξεκάθαρους κανόνες ό,τι αφορά την διασύνδεση ε, και ΕΣΥΦ. Όχι μετά, τώρα λοιπόν, γιατί ήδη τρέχουν τα προγράμματα. Είμαστε λίγοι εδώ σήμερα στην αίθουσα, αλλά αν μιλήσετε με εκπροσώπου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι τη δική σα Γενική Διεύθυνση, από άλλε, αν του ακούσετε λοιπόν, έχουν ε, τον ξεκάθαρο στόχο. Πάρτε χρήματα την πολιτική συνοχή. Δεν θέλω να κατανομάσω κανέναν, αλλά αυτό κάνουν. Γιατί θεωρούν ότι αυτή είναι μια καλή πηγή πόρων που δεν δαπανώνται. Εφόσον δεν δαπανώνται, μπορούμε να τα πάρουμε και να τα διοχετεύσουμε στο ΕΦΣΥ. Όμω, δεν είναι αυτή, αυτός ο σκοπός η αποστολή του έψη. Συμπληρωματικότητα, ναι. Όπως είπατε, ενιαία θηρίδα. κάποιο θέλει να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα. Ποιο πρόγραμμα μπορώ να αξιοποιήσω, ποια κονδύλια, από ποιο ταμείο. Αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε αυτή την πολιτική ε, του κατακαιρματισμού και των στεγανών. Επομένω, συμπερασματικά, α απλουστεύσουμε το σύστημα, ξεκινώντα όμω από την ε, οικοδόμηση εμπιστοσύνη με τους εταίρου. Γιατί δεν γίνεται να υπάρχει ε, απλούστευση χωρί εμπιστοσύνη, είναι ψέμα αυτό. Και όχι blending, αλλά συμπληρωματικότητα. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά. Και βέβαια, η απάντηση θα μπορούσε να είναι Τέλος πάντων, ένα κάτι τελευταίο. Δεν είναι τυχαίο που δύο χρόνια τώρα εργαζόμαστε πάνω στο σύστημα ε, της πολιτικής συνοχής. Στην αρχή της θητείας είχαμε το, τη σύσταση του ΕΦΣΙ. Το σύστημα λοιπόν ήταν έτοιμο. Ο Λάμπερτς ήταν εισηγητής για τον Γενικό Κανονισμό για την Πολιτική Συνοχή και εγώ ήμουνα εισηγητή για το ERDF. Και τελικά ε, βρεθήκαμε με ένα τελείω καινούριο μηχανισμό που μόλις είχε δημιουργηθεί. Έπρεπε λοιπόν να δούμε πόσο ακριβώς θα τα συνδυάσουμε. Τα ξέρετε βέβαια όλα αυτά πολύ καλά. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί έχουμε ακόμα 17-18 μέχρι το 20. Τώρα πρέπει να γίνουν όλα αυτά λοιπόν. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα για να μην έχουμε πολιτική ατζέντα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ χρήσιμο για μας λοιπόν όλα αυτά να τα μεταφράσουμε σε πολύ ε, πρακτικούς όρους και να ξεφύγουμε από το ιδεολογικό και μόνο πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδελφούς που πήραν το λόγο. Ε, νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιον άλλον. Να δώσω λοιπόν τώρα τη δυνατότητα στο πάνελ των πυρογνωμόνων να απαντήσει στις διάφορες ερωτήσεις. Να ξεκινήσουμε αντίστροφα, γιατί νομίζω ότι η πλειοψηφία των ερωτήσεων ε, ήταν ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επομένως θα την αφήσω τελευταία. Να δώσω καταρχάς λοιπόν το λόγο στον κύριο Ουατρί για να πει δύο λόγια. Ε, αν έχετε να πείτε κάτι, ε, τώρα είναι η στιγμή και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Νιούνιος Φεράρ, μετά στον Τσέχο εκπρόσωπο και μετά στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Γουατρί λέγομαι. Όχι βατρί. Εμείς εργαζόμαστε επιτόπου ε, στα προγράμματα των επιχειρήσεων και διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρηματίες ε, παρουσιάζουν κάποια προγράμματα και δυσκολεύονται να αποτανθούν στον κατάλληλο άτομο για να αποζημιωθούν για τις δαπάνες τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε ένα ταμείο επενδύσεων και τους λέμε ότι εμείς έχουμε χρήματα απευθείας τα οποία έρχονται από την Ευρώπη και ε, μπορούμε να σας χρηματοδοτήσουμε αμέσω και αλλάζουν τα πράγματα έτσι. Ε, δεν ξέρω βέβαια από εκεί και πέρα τις ε, διακλαδώσεις και τα θέματα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Αυτό είναι παρατήρηση λοιπόν. Δεν ε, έχω κάτι άλλο να πω επί του θέματος. Ευχαριστούμε κύριε Γουατρή και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Ενούνια Φερέρ. Ελάχιστες παρατηρήσεις έχω να κάνω. Καταρχάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό uh, να αποφύγουμε ε, προβλήματα με την απλοποίηση. Νομίζω ότι ε, στη διαδικασία της ε, απλοποίησης διαπιστώθηκε τα δύο τρίτα των σφαλμάτων προέκυψαν από λανθασμένη ερμηνεία των κανόνων και όχι γιατί κάποιο δεν ήθελε να κάνει τη διαδικασία σωστά. Εξηγήθηκαν και οι λόγοι. Ε, ε, Ορισμένε φορέ υπήρχαν κανόνες που άλλαζαν τους αρχικούς κανόνες. Αυτό είναι το ένα το οποίο ε, προκαλεί αρκετή ζημιά. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να προσέξετε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, εργάζομαι σε ερευνητικά προγράμματα και διάβαζα μία έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για τον ορίζοντα 2020 και έλεγε ότι κάποια Ινστιτούτα δεν μπορούν να ελέγξουν τα ακριβή ποσοστά ε, ε ανθρωπορών ε, και ανθρωποημερών στι οποίε εργάστηκαν και διαπίστωσα ότι κάποιοι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν εργαστεί ποτέ σε ερευνητικό πρόγραμμα. Ορισμένες φορές λοιπόν εγώ εργάζομαι το Σαββατοκύριακο αλλά σε αυτό το ε, πρόγραμμα το οποίο πρέπει να συμπληρώνω τις ώρες μου δεν υπάρχει δυνατότητα να συμπληρώσω το Σαββατοκύριακο. Πού θα τις βάλω. Αν υπάρχει λοιπόν ένα στόχος ε, να υπάρχει ένα προϊόν, να υπάρξει ένα αποτέλεσμα, τότε να ελέγξετε κατά πόσο υλοποιήσετε. Γιατί είμαστε ανταγωνιστικοί προ τι τιμέ. Όταν γίνεται μια πρόταση, ανταγωνιζόμαστε προ τι τιμέ. Το πώ θα χρησιμοποιώ εγώ το χρόνο μου από εκεί και πέρα δεν έχει σημασία και ε, παρόλα αυτά μας υποχρεώνεται να συμπληρώνουμε ένα time sheet που έχουμε τις ε, διάφορες χρονοθυρίδες για το πόσο εργαστήκαμε ενώ το πρόγραμμα είναι ένα καινοτόμα πρόγραμμα και πρέπει να δούμε και τι γίνεται και τι γίνεται αν δεν έχει κάποιο συμπληρώσει τις ώρες εργασίας αυτό δεν αντανακλά την πραγματικότητα. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση δεν έχουν καμία σχέση με το τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί για να επιτύχουν το στόχο τον επέτυχαν ή όχι. Ναι ή όχι. Αν τον πέτυχαν, πλήρωσέ του. Αν όχι, μην του πληρώνει. Αλλά μην δημιουργεί έναν εφιάλτη και μετά το ελεκτικό συνέδριο να λέει ότι πρέπει να ελέγχουμε καλύτερα τι ημέρε εργασία στο πρόγραμμα αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Δημιουργείται επίπλαστη εργασία για επίπλαστους ανθρώπους για να συμπληρώσουν κατ' επίφαση χρονοδιαγράμματα και τελικά αυτό που έχει σημασία να γίνει δουλειά. Και αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα από τα πολλά. Και φυσικά υπάρχουν και λάθη και το ποσοστό σφαλμάτων στη συνέχεια ε, μας δείχνει ότι α, δεν έχει υπογραφεί αυτό και γίνεται ολόκληρη φασαρία γιατί κάποιος ερευνητές ο οποίος ε, βρήκε κάτι δεν συμπλήρωσε τα time sheets αυτά με τις ώρες εργασίας. Κάποιες παρατηρήσεις και από πλευράς μου αρχίζω να χάνομαι στον κόσμο του Ταμείου Στρατηγικής Ανάπτυξης με όλη αυτή τη συζήτηση και πρέπει να πω ότι ε, και εμείς δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς ε, τι διέπει την όλη διαδικασία. Όσον αφορά ε, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει τίποτα όταν έχουμε τελικά απτά αποτελέσματα και θέλουμε να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε για το ΕΦΣΥ και από εκεί και πέρα να αντιδράσουμε από αυτού να δούμε κατά πόσον υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε. Και τίθεται και θέμα και άλλων μέσων, όχι μόνο του Ταμείου Στρατηγικής Ανάπτυξης. Διότι η ερώτηση που πρέπει να τεθεί πριν ε, διαμορφώσουμε το μελλοντικό πλαίσιο είναι γιατί υπάρχουν τόσοι κανόνες και τόσες απαιτήσει όταν είναι συγκεκριμένο ο κατάλογο αυτών που πρέπει να επιτευχθούν. Αν δείτε την πολιτική συνοχή, έχουμε πάμπολου κανόνε. Διαφέρουν τα πράγματα όσον αφορά τους κανόνες και τις απαιτήσει, αλλά από θεματική σκοπιά έχουμε πολλές ομοιότητες. Έχουμε την πρωτοβουλία, για παράδειγμα, για την απασχόληση των νέων και το Connecting Europe Facility, που έχουν συγκεκριμένου στόχου. Επομένω, η ιδέα θα ήταν να δούμε κατά πόσον απλοποίηση ε, μπορεί να σημαίνει και μείωση των πρωτοβουλειών, να υπάρχουν συγκεκριμένε πηγές, ακόμα και μία μεγάλη πηγή. Δεν έχει τόση σημασία. Επίσης έχει σχέση και με τον καθορισμό των συνεργειών και της ε, καθοδήγησης που λαμβάνουμε. λέμε για παράδειγμα, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα στήριξη από αυτό το ταμείο, ας το υποστηρίξουμε από αυτό. Αυτό δεν είναι συνέργεια. συνέργεια είναι να πάρουμε από εδώ και από εκεί και να τα συνδυάσουμε. Ο ορισμός δεν είναι ορισμός συνέργειας στην πραγματικότητα και προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι είναι συνέργεια και τι είναι συμπληρωματικότητα. Και εάν πιάσουμε τον ορισμό, χανόμαστε. μας ενδιαφέρουν οι κανόνες ε, και ορισμένες φορές τα πράγματα γίνονται πολύ περίπλοκα, αλλά ε, απλώς θα πρέπει να τα δούμε λίγο πιο απλοποιημένα και να τα συνδυάσουμε όπως σας έδειξα στην παρουσίασή μου. Μια πολιτική είναι πιο προβεβλημένη όταν μιλάμε με τους πολίτες, όταν είναι απλή. Και αυτό βλέπουμε και όταν συνομιλούμε με τους πολίτες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να απλοποιήσουμε τα πράγματα και να μειώσουμε τα μέσα και να προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε αυστηρά και μόνον στα αποτελέσματα. Για τα σφάλματα τώρα. Αν, δείτε, διαπιστώνετε σφάλματα στην πολιτική συνοχή και τα συγκρίνετε με την έκταση της κατανομής, δεν είναι τόσο μεγάλο το περιθώριο. Μπορούμε να διδαχθούμε από αυτά. Τα πάντα όμως προκαλούνται από πολύ περίπλοκο τεράστιο σύστημα διότι χάνεσαι σε διατάξεις, σε κανόνες που δεν τους κατανοείς, χρειάζεσαι εξηγήσει και είναι τόσοι πολλοί αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται, επομένως σίγουρα θα υπάρξει μια παρανόηση. Πρέπει λοιπόν να διδαχθούμε από όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ωραία. Και για να ολοκληρώσουμε, ο κύριος Βαν Μπρέσκα, εξ ονόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα λίγο να επανέλθω στα όσα είπε ο κύριος Φερνάντης, ο εισηγητής ε, ε, και τα ερωτήματα που έθεσε. Πράγματι στις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης τα κράτη-μέλη ανέφεραν ότι θα αξιοποιήσουν εντό των διαρθρωτικών ταμείων, όχι δηλαδή στο ΕΦΣΥ, διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχουμε για παράδειγμα 24 κράτη-μέλη τα οποία προτίθενται να αξιοποιήσουν 20 δισεκατομμύρια στο πλαίσιο αυτού του, αυτών των ε, μηχανισμών, ε, δηλαδή το διπλάσιο σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Οπότε σας ε, δείχνω εδώ δηλαδή ποια είναι η αναλογία αυτών των ε, χρηματοδοτικών μέσων. Εδώ δηλαδή κάποια, έχουμε να κάνουμε κάποια εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία, άλλα ε, περιφερειακά, άλλα τα οποία είναι υπό την κοινή των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ούτω καθεξής. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα που τέθηκε επανειλημμένα σε ό,τι αφορά το συνδυασμό μεταξύ ΔΕΤ και ΕΦΣΙ στην πρόταση Omnibus. Αυτό που εμείς προτείναμε είναι ένας συνδυασμός στο άρθρο 39 που συνεπάγεται ότι τα κονδύλια αυτά παραμένουν εντός της πολιτικής συνεχής. Δεν δηλαδή εκραίων από αυτόν τον τομέα. Πρόκειται για ένα συνδυασμό μεταξύ ΕΦΣΗ, Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και Διαφθορτικών και Επενδυτικών Ταμείων εθελοντικού χαρακτήρα. Κανένα δηλαδή κράτο μέλο δεν θα είναι υποχρεωμένο να συνδυάσει αυτά τα κονδύλια αν δεν το επιθυμεί. Και επαναλαμβάνω, τα εν λόγω κονδύλια θα παραμένουν εντό του τομέα ε, συνοχής, της πολιτικής συνοχής. Ε, και ε, γιατί θέλουμε λοιπόν να υπάρξει ένα συνδυασμό, πέραν δηλαδή της όλης συζήτηση που γίνεται για τριπλό α και ούτω καθεξής. Επειδή υπάρχουν τόσα πολλά, τόσες πολλές ανάγκες των κρατών μελών, ώστε να μην επαρκούν από μόνα τους τα κονδύλια της, του Ταμείου Συνεχής για να τις καλύψουν. Οπότε, αν μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά τα κονδύλια με τα κονδύλια του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, τόσο το καλύτερο. Γιατί θα πρέπει σε περίπτωση συνδυασμού να έχουμε ένα παράγοντα της τάξης 4. Ε, δηλαδή ε, ο συνδυασμός των κονδυλίων με κονδύλια του ΕΦΣΙ θα πρέπει να ε, σε μία μονάδα αν θέλετε χρηματοδότηση από την πλευρά του ΕΦΣΙ θα πρέπει να προσθέτονται τέσσερις μονάδες εξωγενούς χρηματοδότησης ιδιωτικής και ό,τι καθεξής. Οπότε εάν κάποιο κράτος μέλος επιθυμεί να προβεί σε μία τέτοια αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΦΣΙ ε, και θα είναι θελοντικό, ε, θα πρέπει να διασφαλίζει ακριβώς αυτή την απόδοση σχετικής επένδυσης. Και από εκεί και ε, πέρα, η δημιουργία των χρηματοδοτικών μηχανισμών, η συζήτηση των όρων τους με, τις διάφο- με τους διάφορους χρηματοδοτικούς οργανισμούς της τράπεζας και ούτω καθεξής είναι πολύ περίπλοκο για τους ε, δημοσίους υπαλλήλους. Οπότε, αν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία και όλο το εργατικό δυναμικό, το προσωπικό του ε, που έχει την απαραίτητη την πυρογνωμοσύνη τόσο το καλύτερο. Γιατί βέβαια η όλη συζήτηση πρέπει να γίνεται ε, και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οπότε το να προβαίνει ένα μόνο σε μια επένδυση από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αξιοποιώντα τα όσα μπορεί να προσφέρει το ΕΦΣΥ είναι κάτι το θεμετό. Δεν πρόκειται λοιπόν εδώ στο πλαίσιο αυτής της πρότασης μόνο και μόνο για τον στόχο ε, του να διατηρήσει δηλαδή την αξιολόγηση του τριπλού αλφα Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τώρα εύχομαι στον κανένα 1-3 που αναφέρατε. Ε, ε, σημερινή προγραμματική περίοδο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ακόμα και αν ε, γινόταν μια πρόταση αυτή τη στιγμή από την Επιτροπή, δεν θα γινόταν δεκτή από τα κράτη-μέλη. Γιατί δηλαδή να δεσμευτούν τα κράτη-μέλη ε, ε σε έναν κανόνα πιο περιοριστικό, να πάνε δηλαδή από το 1 3 στο 1 2 ή κάτι άλλο. Το μόνο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση είναι να παρακολουθούμε στενά το τι συμβαίνει, να παρέχουμε υποστήριξη όπου αυτή χρειάζεται, όπου υπάρχουν δηλαδή διοικητικά προβλήματα στο επίπεδο τη εκτέλεση και από εκεί και μετά. Αυτό που ελπίζουμε με βάση και τα, τους αριθμούς ε, δηλαδή επιλογής των σχετικών project να οδηγηθούμε και σε αύξηση των σχετικών δαπανών, των πραγματικών δηλαδή εκταμιεύσεων ε, σε επίπεδο δηλαδή κεντρικού προπολογισμού από τις πλευρά των Πρεξελών. Έτσι λοιπόν αναμένουμε ότι μέσα στο 2017 θα ανταποκριθούμε πράγματι στις εκτιμήσεις που είχαμε κάνει σε ό,τι αφορά την, ε, το ποσοστό εκτέλεση του προπολογισμού. Αφού ακριβώς θα ε, αυξηθεί ο ρυθμό εκτέλεση από το πλευρά των κρατών Πάντω σε αυτήν τη φάση δεν μπορεί να γίνει κάτι ε, περαιτέρω. Από το 2020 και μετά θα πρέπει να ξανασυζητηθεί και πράγματι για μένα αυτή η επιλογή του NC3 ε, αντί για το NC2 ήταν λανθασμένη. Αλλά αυτή είναι δική μου άποψη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι επιδόσει με βάση το output, output based delivery, στην πρόταση Omnibus υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα με φορά αν θέλετε ενό συστήματος σε ένα άλλο πλαίσιο που βασίζεται περισσότερο στο output. Τι σημαίνει αυτό. Εκ των προτέρων συμφωνία σε ό,τι αφορά τους στόχους δηλαδή η καταβολή των ε, πληρωμών γίνεται με βάση ακριβώ την επίτευξη κάποιων στόχων, αλλά ε, τα κράτη-μέλη δεν είναι τόσο ενθουσιώδη. Γιατί? Δεν του ενδιαφέρει τόσο η συμμετοχή. Γιατί? εάν κάποιο ε, αποζημιώνεται με βάση τι ε, δαπάνε τι οποίε έχει καταβάλει, είναι σίγουρο ότι θα λάβει ακριβώ αυτή την αποζημίωση. Αν όμω ε, η καταβολή ακριβώ αυτή του κονδυλίου εξαρτάται από, τον, από την επίτευξη ενό συγκεκριμένου στόχου, μια επίδοση δηλαδή, κάποιο δίκτυο, οτιδήποτε άλλο, υπάρχει ο κίνδυνο να μην λάβει κανεί αυτή τη χρηματοδότηση από την Επιτροπή. Άρα λοιπόν στο μέλλον θα έπρεπε να περάσουμε συνολικά πλέον σε ένα σύστημα το οποίο αντί να βασίζεται στις δαπάνες που προέκυψαν για το πρόγραμμα να βασίζεται στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Ε, ενδεχομένως θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ορισμένες χώρες, σε ορισμένους τομείς, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα τη πολιτική συνοχή. Για παράδειγμα, αν κατασκευάσει κανεί ένα αυτοκινητόδρομο, επειδή ακριβώ θα πρέπει να προβεί στην ε, προκήρυξη διαγωνισμών, θα γνωρίζει ακριβώ το πιο ποιο θα είναι το κόστος για την κατασκευή του. Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ ένα κράτος ε, μέλος ε, να πει ότι ε, εντάξει ας με αποζημιώσει η Επιτροπή για κάθε ε, χιλιόμετρο το οποίο έχει κατασκευαστεί και έχουμε συμφωνήσει 100 χιλιόμετρα. Γιατί αν αυξηθεί για παράδειγμα κατά τη διάρκεια υλοποίηση ε, του project το κόστος για κάθε ένα χιλιόμετρο, τι θα γίνει. Οπότε σίγουρα θα προτιμά το κράτος μέλος να λαμβάνει τη χρηματοδότηση από, το, από την Επιτροπή με βάση τις πραγματικές δαπάνες που προέκυψαν και θα είναι πράγματι ακριβώς αυτό επαληθευόμενε οι δαπάνε αφού όλα θα γινόνται μέσω προκήρυξη διαγωνισμών. Πάντω, σε ορισμένου τομεί και για τα κράτη-μέλη εκείνα που ενδιαφέρονται θα μπορούσε να γίνει αυτή η μετάβαση, αν θέλετε, σε ένα διαφορετικό σύστημα με βάση του στόχου. σω καταρχήν πιλωτικά, δοκιμαστικά, προκειμένου να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να εδρεωθεί ή όχι. Πάντως δεν θεωρώ ότι θα αποτελέσει δηλαδή, αυτή η έμφαση, αν θέλετε, στην επίτευξη στόχων, το όραμα, αν θέλετε, για το μέλλον. Το Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού, πράγματι συμφωνώ μαζί σα. Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη σε όλα τα επίπεδα. Ε, και γιατί έχουμε τόση πολύ καθοδήγηση, τόσο guidance δηλαδή, το οποίο παράγεται. Δεν είναι επειδή εμεί έχουμε μια τέτοια μανία από την πλευρά τη Επιτροπή να προβαίνουμε σε έκδοση κατευθυντήριων γραμμών. Τα κράτη-μέλη μα τη γιατί μα λένε δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε σε δύο-τρία χρόνια από τώρα. Α προετοιμάσει λοιπόν ένα σημείωμα καθοδήγηση ε, η Επιτροπή, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι ακριβώ θα κάνουμε και θα είμαστε εξασφαλισμένοι, αν θέλετε, με αυτόν τον τρόπο. Ε, και βέβαια μετά η μία καθοδήγηση διαδέχεται την άλλη και αυτό βέβαια ε, διαονίζει, αν θέλετε, την έλλειψη εμπιστοσύνη, γιατί τα κράτη-μέλη δεν εμπιστεύονται εμά ω Επιτροπή, εμεί με τη σειρά μα δεν εμπιστευόμαστε τα κράτη-μέλη και Άρα λοιπόν θα πρέπει να επανεξετάσουμε αυτό το σύστημα. Και επίση συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι υπάρχει αλληλεπεκάλυψη μεταξύ των διαφορετικών ε, ε, ταμείων. Εδώ δεν, α, ε, δεν αναφέρομαι μόνο σε επίπεδο ΕΦΣΙ και ΕΣΥΦ, αλλά για παράδειγμα στην διακόνηση συνδέοντα στην Ευρώπη και το Ταμείο Περιφερειακή αλλά και με άλλα ταμεία συμβαίνει το ίδιο. Δηλαδή, ε, μπορεί κανείς να αξιοποιήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ε, ε Ταμείο Ανάπτυξης Υπέθρου, για να χρηματοδοτήσει ουσιαστικά το ίδιο ε, project. Οπότε χρειάζεται μια καλύτερη διαφοροποίηση, οριοθέτηση μεταξύ των ταμείων στο μέλλον και χρειαζόμαστε και μια ενιαία δέσμη κανόνων. Ενδεχομένω και θα πρέπει να συγχωνεύσουμε και κάποια ταμεία. Αλλά βέβαια όλα αυτά είναι πολύ πιο εύκολα στη θεωρία από ό,τι στην πράξη. Για παράδειγμα, το σημαντικό για την Επιτροπή Ζητηματοκρατικών Ενισχύσεων προκύπτει εδώ. Δηλαδή, αν πηγαίνουμε σε κεντρικά ε, διαχειριζόμενα ε, συστήματα, έχουμε ε, ευθύνη, ανάληψη ευθύνη σε επίπεδο κράτους μέλους. Αν έχουμε τώρα κατανομή ε, ανά κράτος ε, μέλος σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση στο πλαίσιο διαφορετικών ταμείων ε, βρισκόμαστε πλέον στον τομέα της κρατικής επιχορήγησης οπότε όλα αυτά πρέπει να περνούν από περαιτέρω ελέγχου. Οπότε αυτό μας οδηγεί στην παράλογη κατάσταση ότι εάν στο Horizon 2020 να μην έχει κανείς την κατάλληλη χρηματοδότηση και πούμε εμείς από την πλευρά της Επιτροπής ότι θέλουμε να το αναλάβουμε εμείς αφού ούτως ή άλλως για το δικαιούχο δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ποιος θα δώσει την ε, χρηματοδότηση. Εάν το κράτο μέλο αποφασίζει μέσω διορθωτικών ταμείων να παράσει τη χρηματοδότηση, θα πρέπει ακριβώ να γίνεται όλο αυτό ο έλεγχο τη συμμόρφωση και ούτω καθεξή. Αυτό όμω είναι ένα γενικότερο ζήτημα που αφορά την πολιτική συνοχή και θα πρέπει ε, βέβαια να το εξετάσουμε και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που επηγάζουν από τι διατάξει τη συνθήκη βέβαια δηλαδή να επιτύχουμε την κατάλληλη ισορροπία, αν θέλετε, μεταξύ των κεντρικά διαχειριζόμενων ε, μηχανισμών και ταμείων και των ε, επιμέρους ταμείων. Τώρα, σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει μια τέτοια αλλαγή η Επιτροπή. Γιατί όπως αναφέρθηκε και επανειλημμένα, εμεί βασιζόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ελεκτικό Συνέδριο για όλα αυτά. Για παράδειγμα, τώρα θέλουμε να περάσουμε στην αρχή του ενιαίου ελέγχου, δηλαδή ξεκινώντα από φέτο το Ελεκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή τη, δηλαδή για την έγκριση τη εκτέλεση του προπολισμού, θα βασίζεται στη δική μας, ε, στις δικές μας εργασίες της Επιτροπής και εμείς με τη σειρά μας βέβαια θα βασιζόμαστε ε, στις εργασίες ε, στα όσα κάνουν τα, κράτη-μέλη. Οπότε εδώ θα πρέπει να εξετάζονται πάντα τα ποσοστά σφαλμάτων, τα οποία βέβαια είναι δυνατόν να αξιολογούνται μόνο σε αιτήσια βάση και μόνο εφόσον ελέγχει κανείς operations όπως λέγονται, δηλαδή συγκεκριμένες δράσεις, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να γνωρίζει αν λειτουργεί κάτι σωστά ή όχι. Όταν όμως αναλογιζόμαστε την απλούστευση αυτή τη στιγμή και λέμε ότι θέλουμε να απαλλαγούμε από τα διαφορετικά επίπεδα ελέγχου, τα τρία επίπεδα ελέγχου, τι θα πρέπει να κάνουμε, γιατί έχουμε το, τον έλεγχο του κράτους μέλους, τον έλεγχο των operations και μετά περαιτέρω έλεγχο σε περίπτωση που εντοπίσουμε ε, κινδύνους. Ε, για παράδειγμα, επενδύσεις που συνδέονται με συγκεκριμένους τύπους κινδύνου. Εάν πούμε λοιπόν ότι θέλουμε να εστιάσουμε μόνο σε δύο από αυτά τα στοιχεία. Ε, στα, ε, δηλαδή στον έλεγχο του συστήματος και στον έλεγχο των κινδύνων ε, και όχι σε κάτι άλλο, τότε δεν θα έχουμε πλέον διαθέσιμα στοιχεία σε ό,τι αφορά τα ποσοστά σφαλμάτων. Και κανένας από εκεί και μετά δεν θα ήταν διατεθειμένος, βέβαια, ούτε το Κοινοβούλιο, ούτε το Ελεκτικό Συνέδριο, να βρεθεί σε μια κατάσταση όπου κανένας δεν θα είναι σε θέση να πει ποια είναι τελικά τα ποσοστά ασφάλματος, ποιε είναι οι παρατυπίες οι οποίε προέκυψαν σε ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμα κι αν ω Επιτροπή θέλουμε να προβούμε σε κάποιε αλλαγέ, θα χρειαστούμε τη σχετική υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελληνικό Συνέδριο, αλλά και φυσικά από την πλευρά των κρατών μελών. Δεν δηλαδή μπορεί να επιληθεί ένα τέτοιο ζήτημα με πρωτοβουλία ε, μόνο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά από την πλευρά μου. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαμπρέσκα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτή η δημόσια κράση και να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Φερνάντες, για να ολοκληρώσει. Και να πω ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ στον Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ τη Γραμματεία και σε όλους εκείνους που βοήθησαν για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης και να ευχαριστήσω και τους εμπειρογνώμονες. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση, η οποία καταδεικνύει ότι χρειαζόμαστε αυτή τη συζήτηση. Όλοι τρέφουμε αμφιβολίες και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα εμπιστευτεί το Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο βεβαίως πρέπει να εμπιστευτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει και τα κράτη-μέλη να εμπιστευτούν τα κράτη-μέλη και να εμπιστεύονται και ο ένας τον άλλον. Είμαστε σε μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή συζητούμε το επόμενο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το FC2, και θα ψηφίσουμε την ε, παράταση του Ταμείου. Θα συζητήσουμε και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ελπίζω να μπορέσουμε να πλουστεύσουμε τα πράγματα, διότι κάθε φορά που αναλαμβάνουμε ένα χαρτοφυλάκιο προσπαθούμε να τα πλουστεύσουμε και μετά απλώς τα περιπλέκουμε τα πράγματα. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η συζήτηση. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή και θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε και σε κάποια συμπεράσματα. Γνωρίζω ότι οι πολίτες χρειάζονται χρηματοδότηση, ταμεία, ανάπτυξη και η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως και ε, ε, το συνειδητοποιώ αυτό. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φερνάντες. Απλώς να ολοκληρώσω λοιπόν και εγώ, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι τροφοδότησαν ε, με τις σκέψεις τους τη συζήτηση, τους συναδέλφους που έκαναν την προσπάθεια να συμμετέχουν σε αυτή την ενδιαφέρουσα συνεδρίαση, αλλά μακρά, και θα ολοκληρώσω ως εξής. Δεν είμαι βέβαιος ότι σήμερα θα λάβουμε τις απαντήσεις, αλλά είμαι βέβαιος ότι θέσαμε τις κατάλληλες ερωτήσεις και ότι ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να ε, τις επεξεργαζόμαστε αν θέλουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα τα οποία θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη. Μου ζητούν εδώ να σας κοινοποιήσω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει 11 Μαΐου Σας ευχαριστώ όλους. Δεν έχω κάτι άλλο να πω για τις εμπειρογνώμονες. Κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πέρασε συνεδρίαση. Oh,